Κυρίε uh, Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καθίστε. Για να μιλήσουμε λίγο για το υπόβαθρο. Φαίνεται ότι το Βέλγιο ή τουλάχιστον το Κοινοβούλιο έχει βρει την ε, μέθοδο εφεύρεση τη σάουνα. Εμεί είμαστε κάπω συνηθισμένοι βέβαια ω Φιλανδία, αλλά πάντω οι θερμοκρασίε που αντιμετωπίζουμε είναι κάπω υψηλότερε από ό,τι συνήθω αντιμετωπίζουμε. Και επιπλέον στη σάουνα την κανονική κάνουμε καμιά βουτιά στην κρύα λίμνη. Άρα μάλλον είναι πιο χαλαρωτικό από αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ. Και μια και έχω και την ευκαιρία προεδρεύοντας σήμερα στην Επιτροπή των Περιφερειών θα σας επισημάνω πως έχουμε εδώ το φυλάδιο της Προεδρίας της προσεχούς, της Φιλανδικής δηλαδή στο Συμβούλιο και σας καλώ να το λάβετε για να ενημερωθείτε και να συμβάλλετε βέβαια αναλόγως και στις εργασίες ε, του επόμενου εξαμήνου. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Εγκρίνεται και σας ευχαριστώ πρακτικά της 134 η Συνόδου Ολομελίας της 10 η και 11 η Απριλίου. Μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και σας ευχαριστώ. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Έχω ορισμένε ανακοινώσει και ω προ αποφάσει αλλά και ενημερωτικέ για δραστηριότητε. Μέχρι σήμερα αλλά και στο εγγύ μέλλον. Καταρχάς, γενικός συζητητής. Πριν αρχίσει η δουλειά της ε, παρός Ολομέλειας, δυνάμει του άρθρου 43 του κανονισμού λειτουργίας ε, η Γενική Συνέλευση, η Ολομέλεια καλείται να εγκρίνει τρεις ε, προτάσεις του Γενικού Εισηγητή. Οι δύο απευθύνονται στη Φινλανδική Προεδρία, στο Συμβούλιο. Η μία φορά. την, ε, τον διορισμό του κυρίου Ανδρέας Ρίπφρο, ως Γενικού Εισηγητή για τις ευφύης πόλεις, νέες προκλήσεις και προσαρμογή στη μετάβαση προς την ουδετερότητα και την τήρηση των στόχων ε, της χιλιετίας στην καθημερινή ζωή. Για τον Οκτώβριο τα έως 9 στην Ολομέλειά μας θα πάει αυτή η έκθεση. Μετά έχουμε την ε, κυρία Κάριελα, έναν γενική εισηγήτρια για την ε, εισήγηση, για την γνωμοδότηση για την ψηφιακή Ευρώπη και λύσεις ανοιχτές προς όλους. Σχέδιο πάλι γνωμοδότησης που θα υποβληθεί απευθεία στην Ολομέλεια της 7ης έως 9ης Οκτωβρίου. Τρίτη πρόταση για το διορισμό του κυρίου Ταντέου Άντρε Τσέλσκι από τη Λιθουανία ως ε, Γενικού Εισηγητή για τη διαμόρφωση της μελλοντική ε, ε, ανατολικής γειτονίας και το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου αυτή τη φορά. Παρακαλώ λοιπόν να εγκρίνουμε την πρόταση, τις προτάσεις αυτές και εγκρίνονται, άρα διορίζονται έτσι οι συγκητές. Η κοινή εκδήλωση για την επέτειο 25 ετών από την ε, σύσταση της ε, Επιτροπής των Περιφερειών και του Κογκρέσου των Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης πριν από 25 χρόνια και έχουν συμβάλει βέβαια σε αυτό το διάστημα στην ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών μια εκδήλωση επαιτειακή και πανηγυρική στο πλαίσιο της Ολομέλειάς μας με τον πρόεδρο Καλ Χάιντ Λάμπερτ, από την Επιτροπή των Περιφερειών και του κυρίου Άντρε Κνάμπε από το Κόγκρεσο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αύριο ξεκινά λοιπόν αυτή η εκδήλωση στι 11.45, 12 παρατέταρτο. Το πρωί θα γίνει η σχετική δήλωση και η πανηγυρική αυτή εκδήλωση θα συνεχιστεί με μια διάσκεψη για την κατάσταση της ε, δημοκρατίας και των τοπικών αρχών στην Ευρώπη το απόγευμα στο κτίριο της Επιτροπής των Περιφερειών και Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής Ζακτελόρ στην αίθουσα 52 για τρεις ώρες. Η εκδήλωση για τις μικρές επιχειρήσεις με φωτογραφική μάλιστα έκθεση και επίση, και στο τελευταίο σημείο της ημερήσια διάταξη, θα έχουμε σήμερα μια εκδήλωση για τις ε, ε, επιχειρήσεις τριών περιφερειών συγκεκριμένα που καλωσορίζω άλλωστε στην Ολομέλειά μας με την απονομή βραβείου ε, για δέκατη χρονιά έχουμε ξεκινήσει το 2011 να απονέμουμε βραβείο στις ε, επιχειρήσεις στις τραμμένες προς το μέλλον με βάση και το in ε, πράξη SPA για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης σας καλώ, σας προσκαλώ σε μια δεξίωση που θα παρουσιάσει ταυτόχρονα και τη φωτογραφία για την, ε, έκθεση φωτογραφίας για το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα κτίρια εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια έκθεση που έχουμε ετοιμάσει, έχουν ετοιμάσει ασκούμενοι κατά τη διάρκεια της ε, πεντάμινης περίοδου ασκήσεώς τους. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη δουλειά που έχουν κάνει για μας και την Ευρώπη ολόκληρη. Ένας διαγωνισμός επίσης ε, για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οργανάθηκε από την πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας ε, της Επιτροπής των Περιφερειών βραβεύθηκαν ε, οι επιλεγέντες ε, μαθητές με τα σχολεία τους, τους απευθύνουμε τα συγχαρητήριά μας και τους περιμένουμε στις Βρυξέλλες. Επίσης για την κατανομή των αρμοδιοτήτων έχουμε μία νέα δημοσίευση σήμερα για την Επιτροπή των Περιφερειών και την κατανομή εξουσιών, όπου καταγράφονται οι εξελίξεις σε σχέση με την αποκέντρωση σε θέματα οικονομικά και δημοσιονομικά σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλη την Ευρώπη και βέβαια την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τον, τον μηχανισμό της επικουρικότητας θα δείτε για το κάθε κράτος σας για να, και θα μπορέσετε και να συγκρίνετε με βάση τα τελευταία στοιχεία που θα βρείτε στο διαδίκτυο την κατανομή των αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Θέμα το οποίο άλλωστε συζητήθηκε και χθε στο Προεδρείο. Πληροφορίες έχετε επίσης στους διαδρόμους έξω από την αίθουσα πιο αναλυτικές. Μπορείτε να ενημερωθείτε περισσότερο για το εργαλείο αυτό και από τον ε, διαδικτυακό τόπο πάλι από, τα, από την τεκμηρίωση που έχουμε έξω από την Ολομέλεια. οι παγκόσμιες ε, τάσεις ε, για το 2030, το εγχείρημα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Στρατηγική και ένα σύστημα ανάλυσης το οποίο μπορείτε να βρείτε σε φυλάδια όπως αυτό που σας δείχνω εδώ στο έδρανά σας αλλά και το πιο ε, αναλυτικό εγχειρίδιο που σας δείχνω τώρα μας ενημερώνουν για τις δραστηριότητες της ΕΣΠΑΣ. Όλα αυτά στη διάθεσή σας και έξω από την αίθουσα παρουσιάζουν τις ε, προκλήσεις και επιλογές για την Ευρώπη. Στα επόμενα χρόνια εντοπίζουν τα πιθανά προβλήματα, τους δυνατούς καταλήτες και τις δυνατότητες για εξέλιξη στο μέλλον. Ευχαριστώ επίσης τον συνάδελφο Βίκτορ Σίγκλ, ελπίζοντας να είναι ήδη στην αίθουσα πρόεδρο του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της Άνω Αυστρίας. και εκπρόσωπο τη Επιτροπή των Περιφερειών τα τελευταία 15, στην Επιτροπή των Περιφερειών τα τελευταία 15 χρόνια, που σήμερα συμμετέχει στην τελευταία του Ολομέλεια. Σα ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε και για την παρουσία σα στο Ελσίνκι στην ΕΣΠΟ πριν από μερικού μήνε, όπου είχαμε και την ευκαιρία με την αντιπροσωπεία σα, την αντιπροσωπεία δηλαδή του Κοινοβουλίου τη Ανώστρια, του τοπικού κοινοβουλίου, να συζητήσουμε διάφορα θέματα και είχατε βέβαια και εσεί την ευκαιρία να επισκεφτείτε διάφορε εγκαταστάσει και να συζητήσετε ζητήματα σχετικά με το μέλλον τη Ευρώπη και θέματα μεθοδολογικά ε, και κατευθύνσεις σχετικές με το έργο των πανεπιστημίων. Σας ευχαριστούμε θερμά. Επίσης ο πρόεδρος της ομάδας Άλντε ενημέρωσε τον πρόεδρο για αλλαγή της ονομασίας της πολιτικής αυτής ομάδας που πλέον ονομάζεται Renew Europe, ανανεώνοντας την Ευρώπη, κατόπιν των αντίστοιχων αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η απόφαση αυτή λαμβάνει ισχύ ευθύ αμέσως. Παρακαλώ τη Γραμματεία να επιληφθεί ώστε να γίνει προσαρμογή σε όλα μας τα έγγραφα. Αυτέ Αυτές ήταν οι πληροφορίες από πλευράς του Προέδρου. Έχουμε τις ε, δηλώσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσω και είμαστε και στην ώρα μας με την έγκριση των γνωμοδοτήσεων με πρώτη αυτή του κυρίου Ντάινε Τούρλαϊς. Παρακαλώ λοιπόν και εσείς και ο εμπειρογνώμων σας να έρθετε στο Προεδρείο. Συγχαίρω δε τον νέο εκλεγέντα δήμαρχο της Ρήγας Τη Λετωνίας με τίτλο τώρα ε, στην έκθεση στην εισήγησή σας «Μακροπεριφερειακές στρατηγικές όπως αυτή για τον Δούναβη, ένα πλαίσιο δεκρατικών συνεργατικών σχηματισμών». Από τη δική μου εμπειρία γνωρίζω πως η Ρήγα, η Λετωνία γενικά ως ένα από τα βαλτικά κράτη, έχει συμβάλει σημαντικά στη στρατηγική τη μακροπεριφερειακή για την Βαλτική αλλά και ιδιαίτερα τελευταία στο πρόγραμμα Interreg και στην ΕΦΗ e εξειδικεύση στην περιοχή της Βαλτικής, η Ρήγα, το Πανεπιστήμιο αλλά και πολλές τοπικές περιφερειακές αρχές έχουν πολύ σημαντική συμβολή στο έργο αυτό. Προσβλέπω λοιπόν στην περαιτέρω συνεργασία τώρα που αναλαμβάνεται και καθήκοντα ως δήμαρχος της Ρήγας. Παρακαλώ, να λάβετε το λόγο. ευρωπαϊκή συνεργατική σχήμα. Ε, και κύριοι, σήμερα εδώ στην Ολομέλεια εξετάζουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησή μου για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές όπως που έχουμε για το Δούναβι είναι ένα πλαίσιο για την προώθηση των διακρατικών συνασπισμών, σχηματισμών. Συγγνώμη. Επίσης, έχουμε και μια δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της μακροπεριφερειακής στρατηγικής της Ένωσης. Ευχαριστώ τη Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου που έθεσε το θέμα αυτό και σε επίπεδο Επιτροπής Περιφερειών αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα και διεθνή φόρουμ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και σε προηγούμενες περιόδους, μία από τις προτεραιότητες της, ε, του επικείμενου νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα είναι η μείωση των ε, περιφερειακών ανισοτήτων. Και αυτή η προτεραιότητα συνδέεται άμεσα με τις μακροπεριφερειακές ε, στρατηγικές, ούτως ώστε τα άτομα που ζουν σε γειτονικές περιφέρειες να έχουν λιγότερες ανισότητες. Έτσι θα συμβάλλουμε στην ανάγκη για συνοχή που αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Δύο έννοιες είναι πολύ σημαντικές σε εμά που είμαστε υπεύθυνοι για την τοπική και περιφερειακή στρατηγική. Η επικουρικότητα και η συνοχή είναι οι πιο ουσιώδεις στόχοι της μακροπεριφερειακής στρατηγικής σε αυτή τη συγκυρία διαπιστώνουμε στην έκθεση της Επιτροπής ότι η συνοχή αυτή μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης δεν έχει ακόμη επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Έχουν αναφερθεί μια σειρά από ζητήματα για την επιτυχή στρατηγική της, ε, την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Βεβαίως ε, υπάρχει ευρεία στήριξη σε όλες τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές για την έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα μπορούσαν να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο, να συμμετέχουν στενότερα στην εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. οι δυνατότητες ε, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν ε, πλήρως εάν δεν έχουν επαρκείς πόρους και προσωπικό όμως οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Πρέπει να επιτευχθεί περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κλαδικών πολιτικών και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Ε, για παράδειγμα, τα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στην 21η Μαΐου για την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών το αναφέρουν. Καλούν, καλούν τις χώρες να δείξουν περισσότερη υπευθυνότητα και να επιτύχουν την κατάλληλη πολιτική στήριξη και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων τοπικών και περιφερειακών φορέων. Επίσης, στη γνωμοδότησή μου αναφέρω ακριβώς αυτό. Επίσης ε, το Συμβούλιο τονίζει ότι όλοι οι φορείς πρέπει ενδεχομένως μέσω δικτύων και προγραμμάτων να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να υπάρχει καλύτερος συνδυασμός πολιτικών και στρατηγικών στις ε, περιοχές προτεραιοτήτων όπως είναι αυτή η κλαδική σχηματισμοί. Έτσι, θα αυξηθεί η συνολική ανταγωνιστικότητα των περιφερειών και της Ένωσης και θα συμβάλλουμε στην κοινωνική, οικονομική και περιφερειακή συνοχή. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε επίσης περισσότερο στην προσπάθεια εισαγωγής οικοσυστημάτων καινοτομίας. Είναι τμήμα της μακροπεριφερειακής στρατηγικής όλα αυτά οι υπεύθυνε ε, γενικές διευθύνσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη, την εσωτερική πολιτική, την επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες πρέπει να συνεργάζονται. Όσοι ε, συμμετέχουν στην προσπάθεια περιφερειακών ε, σχηματισμών μπορούν να προβούν σε ανταλλαγή πρακτικών από χώρα σε χώρα. Επίσης, μπορούμε να έχουμε το μαγικό τρίγωνο ε, την ε, πανεπιστημιακή κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτά θα είναι οι τρεις κορυφές του τριγώνου. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που διαπιστώνω ότι τα περισσότερα, οι περισσότερες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην ε, γνωμοδότησή μου την εμπλουτίζουν. Προτείνω τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες για να καλύψω τις περισσότερες από τις τροπολογίες που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ τη Σουηδική Αντιπροσωπεία για τις ε, προτάσεις της για την πολιτική συνεργατικών σχηματισμών. Βεβαίως δεν θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ αυτών των σχηματισμών πρέπει να περιοριστεί στις περιοχές που καλύπτει η μακροπεριφερειακή στρατηγική. Ευχαριστώ και τη γερμανική αντιπροσωπεία για τις τροπολογίες της για τη δημιουργία νέων μακροπεριφερειακών στρατηγικών και συμφωνώ ότι όταν θα εκπονήσουμε αυτές τις νέες στρατηγικές δεν θα πρέπει να ε, παρακολύσουμε τη λειτουργία των υφισταμένων τέτοιων στρατηγικών. Ευχαριστώ και τους Ιταλούς συναδέλφους για τις προτάσεις τους, για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συνεργατικών σχηματισμών και προτείνω οι δύο τροπολογίες αυτές να ενταχθούν σε μία μόνο παράγραφο γιατί καλύπτουν το ίδιο θέμα. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, τονίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη, όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης μπορούν να είναι τόσο ισχυρέ όσο είναι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος και καθήκον μας είναι να είμαστε ενωμένοι και ισχυροί. Να το έχουμε αυτό υπόψη όταν τώρα εκπονούμε νέες προτάσεις και για τις ε, στρατηγικές μας αυτές και για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλες αυτές τις πολιτικές. Όλα αυτά ε, είναι εντός των δυνατοτήτων μας. Σας παρακαλώ να στηρίξετε την γνωμοδότησή μου μαζί με τις τροπολογίε. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ντάινι Τουρλάι. και να ξεκινήσουμε τη γενική συζήτηση. Γιώζεφ Μπέρενι. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να συγχαρώ τον εισηγητή πολύ καλή βάση γιατί τονίζει ποια είναι τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια που παρεμποδίζουν την ε, επιτυχή εφαρμογή αυτών των στρατηγικών. Είναι οι διαφορές στις διοικητικές δομές. Πολύ σωστά τονίζεται αυτό. Πρέπει να υπερβληθεί αυτή η δυσχέρεια για να εφαρμόσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Κάτι άλλο εξίσου σημαντικό έλλειψη πόρων. Αυτό είναι πάντα το μεγαλύτερο πρόβλημα για να υπάρξουν επιτυχείς στρατηγικές. Αλλά να τονίσω κάτι άλλο. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν παράλληλες δομές και στρατηγικές. Γι' αυτό είμαι υπέρ της τροπολογίας 5 του κυρίου Φλόριαν Σουίτς που λέει ότι αν ήδη υπάρχουν στρατηγικές για κάποιο θέμα δεν θα πρέπει να υπάρξει επικάλυψη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα αλλά και πάλι συγχαίρω τον εισηγητή γιατί είναι πολύ καλό το κείμενό του. Ευχαριστώ. Ο Ρομπέρτο Τζαμπέρτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τι γνώμη έχει για την ε, τροπολογία 3 της ομάδας μου ε, η ε, η οποία νομίζω προτείνει κάτι απολύτως λογικό. Δηλαδή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπορούμε να συγκαταλέξουμε, να συγκαταλέξουμε και την σύγκληση στόχων και τη συνεργασία που θα ενίσχυαν την επιτεύξη των στόχων και θα βελτίωναν και την εδαφική συνοχή μεταξύ των κρατών. Γι' αυτό σας παρακαλώ να αξιολογήσετε το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει. Αυτή η απολύτως λογική για μένα ε, τροπολογία. Okay, thank you. And then, uh, Rafaela... Ευχαριστώ. Ραφαέλα Κατανέο. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεση. και για την ε, έκθεση μάλιστα που ανέλαβε και πριν ε, για το ίδιο θέμα ως ε, πρόσωπος της Επιτροπής. Στο σημείο 3 πάλι θα επιμείνω όπως και ο πρόεδρος Τσαμπέτη καθώς η Ευρωπαϊκή Προεδρία στην ζώνη EU Alpes, Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλπιων δηλαδή που έχει αναλάβει Λομπαρδία ως περιφέρεια Έχουμε μία διάσταση που αφορά την συνοχή για την περιοδο 2021 21-27 και θα θέλαμε μέσα στην έκθεση αυτή, στην εισήγηση αυτή, αλλά και σε άλλες στρατηγικές μακροπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των οποίων και αυτής του Δούναβη, να δώσουμε έμφαση στη συνεργασία αυτή και καλό τον ε, εισηγητή ε, να ε, υποστηρίξει αυτή την τροπολογία την οποία άλλωστε εγώ θα υπερψηφίσω. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία παριθμών 1. Ο συγητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Ουδής εγκρίνεται. 2R, η τροπολογία του εισηγητού, η οποία εφόσον εγκριθεί οι δύο καταπίπτει. Ψηφίζουμε υπέρ κατά εγκρίνεται κανείς δεν ήταν κατά και καταπίπτει υπερθυμών 2 προχωρούμε τώρα α ο εισηγητής θέλει το λόγο παρακαλώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για την τροπολογία παριθμών 3 την οποία σχολίασαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Δεν είμαι ουδόλως αντίθετος ε, στην προσέγγιση αυτής της τροπολογίας, τροπολογίας παριθμών 3, Πρέπει όμως ε, να είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει και τις επόμενες ε, προεδρίες. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος για το κατά πόσον πρέπει να περιοριστούμε εδώ στην ε, συγκεκριμένη προεδρία. Δεν ήθελα εγώ να υπερβώ ε, τα όρια μου ε, και την εντολή αν θέλετε, αλλά δεν είναι ότι και είμαι αντίθετο. Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ της τροπολογίας. κατά. Κάποιοι είναι κατά, οι περισσότεροι όμως είναι υπέρ, οπότε εγκρίνεται η τροπολογία και προχωρούμε στην τροπολογία 4 του εισηγητή που αν εγκριθεί ε, θα οδηγήσει στο να καταπέσουν οι τροπολογίες 4 και 5. Βράντισλαβ Όρτιλ, ε, παρακαλώ, έχεις ζητήσει το λόγο, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να στηρίξω τη συμβαστική τροπολογία 4R του εισηγητού. Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμιστεί το εξή. Η Επιτροπή μα είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία θέλει να ε, θεσπιστούν νέε τέτοιε μακροπεριφερειακέ στρατηγικέ που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη των ε, περιφερειών. Είναι σημαντικό ε, στην τροπολογία αυτή να σημειώσουμε πως δεν θα πρέπει να περιπλέκει ε, ήδη υφιστάμενες στρατηγικές. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μειωθεί η χρηματοδότηση για παράδειγμα των ήδη υφιστάμενων ούτε να υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις. Η διαχωριστική γραμμή για τη χρήση ευρωπαϊκών κονδύλων είναι γνωστή, είναι σαφής Άρα νομίζω ότι πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση η τροπολογία 4 και θα τη στηρίξουμε ως συμβιβαστική πρόταση. Πρόεδρος, ωραία. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική τροπολογία 4R της ηγητού. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Κανείς εγκρίνεται. 4 και 5 καταπίπτουν. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 6. Ο είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 7 άρτηση γητού αν εγκριθεί καταπίπτουν οι 7 και οι 8. Ψήφι υπέρ τη συμβασία τροπολογία του εισηγητού υπέρ. Κατά. Κάποιοι. Αλλά οι περισσότεροι έχουν ψηφίσει υπέρ. Άρα εγκρίνεται η 7R. Καταπίπτουν οι 7 και 8. Τροπολογία 9 του εισηγητού. Αν εγκριθεί, καταπίπτουν οι 9 και 11. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ, τη 9. Ευχαριστώ. Κατά. Α, εγκρίνεται γιατί δεν υπήρχε καμία ψήφι. Κατά και καταπίπτουν οι 9 και 11. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται. 11. Όχι κατέπεσε. 12. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Κανείς αποχές. Καμία. Ομόφωνα εγκρίνεται η γνωμοδότηση του κυρίου Τουρλάης. Συγχαρητήρια. Uh, Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη γνωμοδότηση του Κριστόφ Ρουγιό. Να έρθει παρακαλώ ο κύριος Ρουγιό στο βήμα με τον εμπειρογνώμονα του και τον εκπρόσωπο της ΕΚΟΝ προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το αντικείμενο της γνωμοδότησης. Έχουμε και εδώ κάποιες τροπολογίες. 16 συνολικά έχουν κατατεθεί και όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση θα τις θέσω σε ψηφοφορία το ίδιο και ορισμένες τροπολογίες του εισηγητού. Κριστόφ Ρουγιό, έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αντιλαμβάνομαι πως το σχέδιο γνωμοδότησης που σας υποβάλλω σήμερα από πολιτικής πλευράς είναι επίμαχο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ούτε από ιδεολογικής ε, ε, πλευράς και πολιτικής ούτε από εθνικής πλευράς μεροληπτεί αυτή η έκθεση. Νομίζω ότι συμφωνεί άλλωστε και με την κοινή γνώμη και τις απόψεις της, διότι με βάση το ευρωβοβαρόμτρο περίπου 75% των Ευρωπαίων θεωρούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη δράση ε, για, τον, ε, για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροαπάτης. Το ίδιο ε, και με την ανάγκη καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής ε, και για μια πιο δίκαιη φορολογία, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκά κινήματα σχετικά. Το ίδιο ε, πιστεύουν και οι μεγάλες πολιτικές οικογένειες, το είδαμε και στις ευρωεκλογές, το ΕΛΚ, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι πράσινοι. Ιδίω η ε, επικεφαλής ψηφοδελτίων, ε, Spitzenkandidat, δε ιδίω του ΕΛΚ, Γερμανό ε, στην εθνικότητα, είπε πω η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λαμβάνει περισσότερε αποφάσει με ειδική πλειοψηφία και στην επόμενη θητεία επιτέλου θα πρέπει η GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple να πληρώνουν δίκαια, δίκαιου φόρου, να φορολογούνται δίκαια το και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κληροδότημα του Ζαν Κλοντ Ιουνκέρ, ξέχοντας προσώπου της οικογένεια του ΕΛΚ, ο οποίο και κατέθεσε την αρχική πρόταση και τη συμπεριέλαβε στα πέντε βασικά ζητήματα για το μέλλον. Ο κύριος Γιούνκερ μίλησε για την ανάγκη μιας δίκαιης σύγχρονης φορολόγησης που θα είναι προσαρμοσμένη στις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας που θα εξασφαλίζει ισότιμη συνθήκες για πλατφόρμες ηλεκτρονικές, για τοπικές επιχειρήσεις και λοιπούς ε, παράγοντες αγοράς. 21 Ιουνίου οι Αρχική κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν και την ε, στρατηγική που κάνει λόγο για την πρόοδο προς μια δίκαιη αποτελεσματική ευρωπαϊκή φορολογία. Ελπίζω λοιπόν πως οι συντάκτες των τροπολογιών και ιδίως ο συνάδελφος και φίλος Μέρφυ θα συμφωνήσουν στη σημερινή ψηφοφορία με αυτά που πρεσβεύει η ηγεσία ε, του ΕΛΚ, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Κομισιόν και της Κοινής Νόμης και τουλάχιστον ε, ιδίω μάλλον τροπολογία 1, θα, θα απορριφθεί αυτομάτως. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου θα ήθελα γρήγορα γρήγορα να σας μιλήσω για τέσσερα θέματα. Πρώτον ανταγωνισμός, δεύτερον κυριαρχία, τρίτον επικουρικότητα, τέταρτον δημόσιες υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, ναι, είναι απαραίτητος ανταγωνισμό ανταγωνισμός για τη λειτουργία μιας κοινωνικής οικονομίας τη αγορά. Δεν είμαστε αφελεί. Γνωρίζουμε πως ε, η τοπική αυτοδιοίκηση επίσης ε, προσφεύγει στο φορολογικό ε, ανταγωνισμό που θα πρέπει όμω να είναι ισότιμος αφορτιόρι σε έναν εναρμονισμένο οικονομικό χώρο σε ό,τι αφορά τους κανόνες που ισχύουν για την εσωτερική αγορά, τις κρατικές ενισχύσεις ή τη μακροοικονομική διακυβέρνηση η ευρωπαϊκή φορολογία δεν θα πρέπει να γίνει ο αδύναμος κρίκος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σε αυτό το κοινό οικονομικό χώρο και ιδίως στην Ευρωζώνη πλέον δεν μπορεί κανείς να φανταστεί η ευρωπαϊκή πολιτική να ε, είναι ε, απλά ένα άθροισμα των εθνικών πολιτικών. Ε, πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε για να πετύχει το ευρώ πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους κοινή οικονομικής ε, πειθαρχία ε, και για μία αν θέλετε συγχώνευση των ε, κυριαρχών η φορολογική κυριαρχία των ΜΕΝ ολοκληρώνεται εκεί που αρχίζει η φορολογική κυριαρχία των ΔΕ όπως θα έλεγε ίσως η Ρόζα Λούξεμπουργκ η πρόταση τώρα της Κομισιόν μιλάω για την κυριαρχία δεν θέλει να δώσει νέες αρμοδιότητες δεν αποσκόπησε να δώσει νέες αρμοδιότητες στην Ένωση ούτε στόχος της Κομισιόν να περιορίσει τις προνομίες των κρατών μελών είναι να σε οτι αφορα τον καθορισμο των συντελεστων αμεση φορολογηση φυσικων προσωπων η επιχειρησεων επομενω η προταση τη Κομισιόν συνάδει απόλυτα με την αρχή της επικουρικότητας. Τέλος, για να μιλήσω για την ίδια την αρχή του φόρου. Δεν είναι κάτι δημοφιλέ σίγουρα οι φόροι, αλλά χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ότι μόνο τα φορολογικά έσοδα τα οποία σπράττονται με αποτελεσματικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη, στι ε, τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ και ε, στα κράτη τελικά να παρέχουν ικανοποιητικέ υπηρεσίε στον τομέα τη παιδεία, τη υγεία, τη στέγαση, τη ασφάλεια, τη καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, τη χρηματοδότηση και τη εφαρμογή των στόχων Βιώσιμη λοιπόν βιώσιμης ανάπτυξης. Συντομία, όταν θα ψηφίσετε, να έχετε στο νου σας ε, την έννοια φορολογία, αλλά όχι ε, ως προς ε, τα συμφέροντα της Amazon και της Apple, που δεν δημιουργούν παρά ελάχιστες εργασίας στην Ευρώπη και μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνες τους, πολύ καλά. Αλλά σκεφτείτε τι γίνεται με τον παντοπόλη της γειτονιάς σας, το φούρναρι, το βιβλιοπόλη, τις δημόσιες υπηρεσίες, και την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν οι δημόσιες επενδύσεις σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Α, παρακαλώ. Ο κύριος Γιώκμαν. Ναι, συγγνώμη, αλλά πρέπει να παρέμβουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρά τι ε, προσπάθειε που κάναμε, δυστυχώ η ομάδα μου, το ECA, δεν μπορεί να στηρίξει αυτήν την γνωμοδότηση για μια σειρά από λόγου. Εάν δεν εγκριθούν οι τροπολογίε 11, 14 και 15, δυστυχώ ε, δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Θεωρούμε ότι η φορολογική πολιτική και η αρμοδιότητα επιβολής φόρων είναι κυρίως θέμα εθνικής κυριαρχίας. Δεν μπορεί να ισχύει ένας κανόνας για όλους. Κάθε χώρα έχει την οικονομική της κατάσταση και ε, τα φορολογικά μέσα είναι ουσιώδη για την οικονομική διακυβέρνηση. Δεν θεωρούμε ότι η εισαγωγή της ε, ειδική πλειοψηφία για, για φορολογικά θέματα θα οδηγήσει σε καλύτερη νομοθεσία. Αντίθετα, θα γίνει κατάχρηση εξουσιών που δεν θα σέβονται πλήρω το δικαίωμα των κρατών μελών να ασκούν τη φορολογική του πολιτική. Επίση, θεωρούμε ότι ο φορολογικό ανταγωνισμό ωφελεί την ενιαία αγορά γιατί ασκεί πίεση από των κρατών μελών για να έχουν μια αποτελεσματική φορολογική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανένα άλλο το λόγο. Όχι. Να ψηφίσουμε. Α, παρακαλώ εσείς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για να, κάνουμε περισσότερη, για να φτιάξουμε περισσότερη Ευρώπη, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, όχι, λιγότερο, όχι λιγότερη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που ισχυρίζονται οι συνάδελφοι του ECR. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το να ξεφύγουμε από το κανόνα της ομοφωνίας μας οδηγεί στο δρόμο προς την περισσότερη Ευρώπη. Έχουμε μια διαδικασία αποφασιστική, λήψη αποφάσεων πολύ πιο δημοκρατική και ισότιμη. Εάν περάσουν οι τροπολογίες του ECR και όχι μόνο μία του Μέρφυ, πηγαίνουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όχι προς την περισσότερη Ευρώπη, αλλά ο δρόμο μας σε σχέση με αυτή και γι' αυτό δεν μπορεί η Επιτροπή των Περιφερειών λάβουν τέτοια απόφαση ε, κάνοντας επιλογές που θα ήταν εις βάρος του, ε, του ρόλου και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σύνορα η Ευρώπη δεν έχει τα σύνορα τα έχουν, το web μάλλον δεν έχει τα σύνορα τα ορίζουν τα κράτη το web, το ίντερνετ έχει το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο μέσα και πρέπει να δώσουμε απαντήσεις ουσιαστικές στους πολίτες μας αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας χωρίς να κοιτάμε τα δικά μας ιδιαίτερα συμφέροντα που μπορεί σήμερα να τα συμφέροντα του ενός κράτους μόνο και όχι των υπόλοιπων, όχι όλων των κρατών. Έτσι λοιπόν η δική μας ευθύνη είναι να κάνουμε περισσότερη Ευρώπη. Η δική μας συμπληρωματικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρώπης ολόκληρης είναι να μπορέσουμε και εκεί θα κρυθεί και η επιτυχία μας να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα οποία αφορούν, απασχολούν την κοινή γνώμη προς το συμφέρον της κοινή γνώμης και ιδιαίτερα για μας που είμαστε τοπικοί άρχοντες και εκπρόσωποι είναι καθήκον αυτό ηθικό, είναι υποχρέωση και αποστολή και γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την τροπολογία στην ουσία και την ε, τροπολογία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μιλάνα. Παρακαλώ για να απαντήσετε κύριο Φιό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Από την προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής μας η προσπάθειά μας ήταν να βρούμε συμβιβαστικέ λύσεις, να διευκρινίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και δεν θέλουμε καμία τροποποίηση της κατανομής αρμοδιοτήτων ή των κανόνων λήψη αποφάσεων όπως αυτοί ισχύουν τώρα και γι' αυτό και δέχθηκα τις τροπολογίες ε, του συναδέλφου Φονρές και μάλιστα υπενθυμίσαμε ξεκάθαρα πώς ε, στηρίζουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, θέλω να τονίσω πώς ε, επιτέλους δίνεται μια απάντηση και στις προσδοκίες των πολιτών. Δηλαδή, βάζουμε ένα τέρμα στο, στην άγρια δύση τη φορολογική που διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί το Amazon να ορίζει ποιοι κανόνες θα ισχύουν και με ποιους όρους μέσα σε ένα κράτο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε τι περιμένει η κοινή γνώμη. Βεβαίω ε, μπορεί κανεί να πει Α, δεν χρειάζεται να κοιτάμε τι θα πούνε οι πολίτε. Εμεί αυτό ω ε, ε, τοπικοί και περιφερειακοί πρόσωποι το ξέρουμε. Αλλά πρέπει να δούμε και τι θα πούνε οι πολίτε στην ώρα των εκλογών. Αυτή τη στιγμή πρέπει λοιπόν να μπει χρήμα στον δημόσιο κορφανά που θα χρηματοδοτήσει και τι δικέ μα τι τοπικέ περιφερειακέ αρχέ. Χωρί να προτείνουμε κάτι το επαναστατικό, νομίζω ότι απλώ τακτοποιούμε τα πράγματα. Βάζουμε μια σειρά στο κατάστημα θα πω ε, με πολιτικές οι οποίες αποβαίνουν σ' όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε. Τροπολογίες 1 15 που έχουν τον ίδιο στόχο και το ίδιο περιεχόμενο. Ας τις δούμε λοιπόν πρώτες και ξεκινώ υπέρ της, ε, των τροπολογιών 1 και 15. Παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Το ναι υπέρ της τροπολογίας, το όχι κατά. Okay, we close the vote. Πέρας απερίφθη σαν πλειοψηφία κατά τροπολογία 2 ρότου εισηγητή για να καταπέσει η 3 εάν εγκριθεί ψηφίζουμε παρακαλώ κατά ηλεκτρονικά πάλι Πέρας. Εγκρίνεται. Οι δύο και οι τρία λοιπόν καταπίπτουν. Πάμε στο συστήν 4. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Όχι. Παρακαλώ. Πρόεδρε, είναι πολύ πολύ βραδύ το μηχάνημα που μου έχουν δώσει. Καλώς, καλώς. Επειδή πατήσαμε το κλειδί ότι έκλεισε, ε, ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε πάλι την τροπολογία υπαριθμών 4 παρακαλώ, ναι ή όχι. Μου λέει ότι κάνει αποστολή, Πρόεδρε, αλλά δεν έχει σταματήσει. Καλώς, περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε μέχρι να έρθει και το δικό σας αποτέλεσμα. Δούλεψε τώρα, εντάξει. Ναι, βλέπω ότι καταγράφονται περισσότερες ψήφοι από ό,τι πριν. Ψηφίσατε όλοι πλέον. Πέρας. και η πλειοψηφία είναι υπέρ. Επομένως εγκρίνεται υπαριθμόν 5. Ψηφίζουμε παρακαλώ υπέρ. Να κάνουμε ηλεκτρονικά. Ah, uh, Όχι. Διανατάσσεως λοιπόν υπέρ. Είμαστε στην τροπολογία 5. Υπέρ της τροπολογίας υπαριθμών 5 παρακαλώ. Κατά. Ωραία. Απερίφθη. Υπαριθμών 6. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά. Have Ψηφίσατε όλοι. Όχι ακόμα. Περιμένουμε. Εντάξει τώρα ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Η πλειοψηφία κατεψήφισε. Περίφθη λοιπόν. Επτά ρο του εισηγητή Εάν εγκριθεί καταπίπτουν οι 7, 8 και 9. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Οι 7, 8, 9 καταπίπτουν. Οι 10. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται υπαριθμών 11 η οποία εγκρινόμενη οδηγεί σε καταπτώση 12 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 υπέρ κατά Απερίφθη. 14 υπέρ κατά Απερίφθη. τη 15 την έχουμε ήδη ψηφίσει 16 παρακαλώ υπέρ κατά ηλεκτρονικά τη 16 All have voted now. Ψηφίσατε όλοι. Όχι ακόμη. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Εντάξει, μπορούμε να κλείσουμε τώρα την ψηφοφορία. Απορρίπτεται με μικρή πλειοψηφία. Και τώρα τελική ψηφοφορία για την τροποποιηθή σαγνωμοδότηση. Υπέρ παρακαλώ κατά εγκρίνεται αποχές εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η γνωμοδότηση αυτή και συγχαρητήρια Let's λοιπόν, επόμενη γνωμοδότηση. Η συγκίτρια Τσονέτ Μάγιο. Μία προσέγγιση της στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να βασίζεται, που να έχει την τοπική διάσταση στο κέντρο της και τονίζω ότι μόλις έρθει ο Επίτροπος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Κατάινεν θα συνεχίσουμε τη συζήτηση ψηφοφορία, σε όποια φάση βρισκόμαστε για να κάνουμε τη συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν. Okay. Okay, here. Οπότε, δυστυχώς η κυρία Μπαγιό δεν μπόρεσε να έρθει μαζί μας και την αντικαθιστά ο κύριος Χέρτερ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, έχετε την γνωμοδότηση για μια βιομηχανική πολιτική της Ένωσης που να βασίζεται στην περιφερειακή και τοπική διάσταση. Αυτό γίνεται μόνο εάν δημιουργήσουμε καινοτόμα οικοσυστήματα και αν συνεργάζονται οι περιφέρειες μεταξύ τους σε δέσμες πολιτικών. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τοπική πολιτική για να έχουμε καλύτερες καινοτομίε και να συνεργαζόμεθα καλύτερα με περισσότερες και άλλες περιφέρειες. Μόνο έτσι θα ενισχυθούν οι περιφέρειες και ο μηχανικός κλάδος. Οπότε η οικονομία συνολικότερα, οπότε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση τη ψηφιοποίηση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης. Χρειαζόμαστε ισχυρές περιφέρειες που θα έχουν επίπτωση και στις άλλες, στις όμορες περιοχές. Όσο, ισχυρή είναι, όσο πιο ισχυρή είναι μια περιοχή, τόσο πιο πολύ βοηθάει τις όμορες. Το Ίντερεγ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει, οπωσδήποτε, αυτή η διαπεριφερειακή συνεργασία να στοχεύει στην καινοτομία και στην εξειδίκευση Όλα αυτά συντονισμένα για να μαθαίνουν η μένα από τα λάθη των άλλων. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Right. Uh, Οπότε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Θέλει κανείς άλλο το λόγο? Όχι. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία του εισηγητή 2R υπέρ παρακαλώ. Κατά εγκρίνεται. Καταπίπτει 2. Τροπολογία 3. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά που εγκρίνεται τροπολογία. Α, παρακαλώ, ο κύριος Μπορ. Ένα έτοιμα παρακαλώ. Η τροπολογία μπορεί να είναι ε, χωριστή παράγραφος. Να μην ε, ενταχθεί στην ήδη υπάρχουσα παράγραφο για το σημείο αυτό. Εντάξει, καλώς. Συμφωνεί ο εισηγητής. θα εισαχθεί ως χωριστό σημείο. Μετά το σημείο 2, μάλιστα. Να το ψηφίσουμε όμως παρόλα αυτά και αυτό υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Κανείς, εγκρίνεται. Λοιπόν, να ψηφίσουμε από κοινού τις τροπολογίες 5, 6 και 7. Από κοινού λοιπόν, υπέρ παρακαλώ κατά μία ψήφος κατά εγκρίνεται λοιπόν 8 ο συγητής κύριε πρόεδρε αυτή η τροπολογία αφορά ένα και μόνο τομέα και δημιουργεί φραγμούς στο εμπόριο και αύξηση του κόστους. Ενώ ο στόχος μας είναι μια συνολική βιομηχανική πολιτική. Η τροπολογία αυτή ε, περισσότερο θα είχε θέση σε μια γνωμοδότηση για ορισμένους συγκεκριμένους τομείς του διεθνούς εμπορίου. Είμαι λοιπόν κατά. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, η τροπολογία αφορά ένα συγκεκριμένο τομέα, αλλά έχει τον ίδιο στόχο με την επίτευξη δηλαδή του 20% συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ. Και ο Χάλιβας είναι πολύ σημαντικό τμήμα του βιομηχανικού μας ε, πυρήνα λόγω της, της, των χαμηλών τιμών των εισαγωγών έχουμε υπερβολικό δυναμικό στην ε, Ένωση. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια έναντι σε αυτό το παράδοξο. Οι χαλιβουργίες μας που πάνε σε τρίτες χώρες για να βρουν πιο ευνοϊκές συνθήκες λειτουργίας δεν θα, δεν θα προκαλέσουν εκεί λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα ανατόνο χάλιβα Μειώνουμε έτσι τις εκπομπές της Ευρώπης, αλλά αυξάνουμε τις εκπομπές μέσω των προϊόντων που εισάγει η Ευρώπη. Χρειάζονται λοιπόν περιβαλλοντικοί δασμοί για να υπάρχουν οι ίδιοι περιορισμοί για τα προϊόντα αυτά με αυτά τα οποία ε, υφίστανται στην Ευρώπη. Ε, γιατί στην ουσία λοιπόν ε, εισάγουμε διοξείδιο του άνθρακα και χάνουμε απασχόληση. Ωραία, θα ψηφίσουμε από αυτού. Ο είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Μα οι περισσότεροι δεν ψηφίσατε. Μα ρωτήσατε δύο φορές ψηφίζουν κατά. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Uh, κατά. Η πλειοψηφία είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Υπέρ η πλειονότητα. Τροπολογία 10. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Κάποιοι κατά, αλλά εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ο συγητή είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία του συγητη 12 12R. Αν εγκριθεί, καταπίπτουν οι 12 και 13. Υπέρ παρακαλώ τις τροπολογίες του συγητή, Ευχαριστώ κατά. Κανείς. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν οι 12 και οι 13. Από κοινού ψήφιση των 14, 15, 16 και 17. Υπέρ παρακαλώ και για τις 4. Ευχαριστώ κατά κανείς. Εγκρίνεται. Τροπολογία του εισηγητή 18R. Εάν εγκριθεί καταπίπτει 18. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά κανείς. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 18. Από κοινού ψήφιση. Από την 19 μέχρι την 28. Εντάξει. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Κανείς. Εγκρίνονται. Τροπολογία του συγητή 29α. Αν εγκριθεί, καταπίπτεται 29. Ποιοι είναι υπέρ τροπολογίας του συγητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Η πλειονότητα είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Ο συγητής είναι κατά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως, η τροπολογία αυτή, η 30, πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος σε πλαίσια οικολογικής αλλαγής. Εάν επεκτείνουμε την κατάσταση και στην, την ε, εξέταση και στη Γεωργία, αποδυναμώνουμε αυτή την προσπάθεια. Ωραία, ο εισηγητής είναι κατά. Ε, ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κατά. Περισσότερο είναι υπέρ. Εγκρίνεται από κοινού ψήφιση 31 έως 34. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί. Ωραία. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Κανείς. Εγκρίνονται. Τροπολογία του εισηγητή 35R. Αν εγκριθεί, καταπίπτει 35. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Λοιπόν, για να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Can we not yet? Okay, keep on sending. Can we now close the... Μπορούμε τώρα να κλείσουμε την ψηφοφορία. Ωραία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε την τροποποιηθήσα τώρα γνώμοδότηση υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Όχι. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστούμε τον κύριο εισηγητή. Και παρακαλώ μεταβιβάστε και στην κυρία Σιγιόν. Uh, Προχωρούμε στο ψήφισμα, που είναι το επόμενο σημείο, με θέμα προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για τη νέα νομοθετική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση, αλλά όπως είπα θα διακόψουμε και θα συνεχίσουμε μετά. Ε, θα διακόψουμε άμα τη αφήξει του Αντιπρόεδρο κ. Κατάινεν. Λοιπόν, ο κύριος Κάιζερ είναι ο πρώτος που θα λάβει το λόγο. Uh, Mr. Kaiser. Mr. Kaiser, είστε εδώ. Excuse me, but I will... Συγγνώμη, αλλά εγώ το λόγο δεν τον θέλω για αυτό το θέμα, αλλά για την συζήτηση με τον κύριο Επίτροπο. Άντρος Καραγιάννης τότε. We seem to have the false You want to go? Κύριε Καραγιάννη, θέλετε το λόγο. Πρόεδρε, απλώς διαβάζοντα ε, τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα νομοθετική περίοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διάβασα ότι γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα Εράσμου για του τοπικού και περιφερειακού εκπροσώπου. Θεωρώ ότι χρειάζεται αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε, γιατί εμεί οι εκπροσώποι τη τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν, δεν τα γνωρίζουμε όλα. Για να προωθούμε και τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γνωρίζει και ο κόσμος τα ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει και τη λειτουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Ήδη κάποια προγράμματα που διοργανώνονται, όπως το Europe for Citizens ή ο διάλογος με τους Ευρωπαίους πολίτες, δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Όμως, επαναλαμβάνω ότι και εμείς ήδη στην τοπική αυτοδιοίκηση χρειαζόμαστε επιμόρφωση για να προβάλλουμε τις θέσεις και τις αξίες και την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιούρα Βρόμπα. Uh, let me please, uh, declare the position. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το ψήσμα για την περίοδο 2019-2024. Εγώ εκπροσωπώ την ομάδα του ECR αυτή τη στιγμή. Στο ψήφισμα αναφέρονται κάποιοι στόχοι που στηρίζει η πολιτική μα οικογένεια, ανευτικό δυναμικό να ανανεωθεί, να υπάρξει φορολογική ε, αναταξινόμηση, η εδαφική συνοχή, μελέτη αντικτύπου τη νομοθεσία για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και ανάγκη για μελέτε ε, εδαφικού αντικτύπου για όλα τα νομοθετικά θέματα. Όλα αυτά είναι θετικά έχουμε καταθέσει δύο, ε, έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίες που δεν ε, μας βρίσκουν σύμφωνους για την ε, ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για τα φορολογικά στο Συμβούλιο και για την κοινωνική πολιτική. 7 και 17 είναι οι δύο τροπολογίες αυτές. Είναι κόκκινη γραμμή για τη δική μας πολιτική ομάδα. Όλα αυτά ε, σχετίζονται με την εθνική κυριαρχία και δεν συμφωνούμε με την υπόθεση ότι με την ψηφοφορία των θεμάτων των κοινωνικών και των φορολογικών με ειδική ε, πλειοψηφία ε, δεν θα οδηγήσει τελικά την, τον αποκλεισμό των μικρότερων. Αντίθετα και θα αποκλείσει μικρότερες χώρες και θα υποβαθμίσει τη δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών, εμείς θα συνεχίσουμε να έχουμε μια σημαντική θέση στην νέα Ευρωβουλή και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε τις προτεραιότητες μας. 62 μέλη από 15 κράτη ε, μέλη θα έχουμε. Κάτι σημαντικό για μένα είναι ότι οι εκλογές έδειξαν πως ε, δεν κατάφεραν να σημειώσουν τόσο υψηλά ποσοστά οι ακραίοι. Σχεδόν δεν έχουμε ε, ακροδεξιούς ε, πολιτικούς. Ε, στη Σλοβακία, τη χώρα μου, δύο ακραίοι εξελέγησαν. Ο Γιάννη Ζαχράντιλ, Σπίτσεν Καντιντάτα, είναι ο πρώτος από την Κεντροανατολική Ευρώπη και του εύχομαι κάθε επιτυχία, όπως και στους υπόλοιπου συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βαν Ράις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πιο γενικόλογος ε, στην προσέγγιση μου. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πολύ ε, που θα υπάρξει μια ψηφοφορία γιατί θυμάστε ίσως ε, τι πανικός επικράτησε μετά την ψηφοφορία το Brexit και θα θυμάστε ενδεχομένω ε, και το χάσμα το οποίο διευρύνθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών της Ένωσης. Εμείς ε, όλες οι επιτροπές ε, συμφωνήσαμε και καταρτήσαμε ένα πολύ σαφές ε, κείμενο. Μεταφέρουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δικές μας προτεραιότητες. Άλλωστε είμαστε αυτοί που είμαστε πιο κοντά στους Ευρωπαίους Πόλεις από θεσμικής πλευράς, ε, δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες. Και ελπίζω ότι στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο θα τοποθετούμαστε γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταδείξουμε στον Ευρωπαίο πολίτη ότι ασχολείται με τα θέματα του Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να παρακολουθούνται δραστηριότητε μας ε, του σύνοικης. Okay. Thank you. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις αυτές και να περάσουμε παρακαλώ στην ψηφοφορία. Uh, amendment number one. Τροπολογία 1. Ψήφι περ. Κατά κανείς εγκρίνεται. Έχουμε μία προφορική συμβιβαστική τροπολογία που συνδυάζει τις τροπολογίες 2 και 4. Τη βλέπετε στην οθόνη την πρόταση, την προφορική αυτή. Ελπίζω να τη διαβάσατε όλες και όλοι. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται. Καταπίπτει τροπολογία παρθυμών 3. Προχωρούμε στην τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται προφορική συμβιβαστική για την τροπολογία 6 στην οθόνη σας. Παρακαλώ, θα τη δείτε. Να ψηφίσουμε λοιπόν ψήφι υπέρ της προφορικής συμβιβαστικής τροπολογίας. Ποιοι είναι κατά, λίγοι. Η πλειοψηφία είναι υπέρ, επομένως εγκρίνεται και καταπίπτει η αρχική τροπολογία 6. Τροπολογία 7. που συμφωνεί και με την γνωμοδότηση Ρουγιό. Ψήφι υπέρ. Κατά. Να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Μπορούμε να κλείσουμε παρακαλώ. Την ψηφοφορία έληξε λοιπόν η ψηφοφορία και η πλειοψηφία είναι υπέρ, εγκρίνεται η συγκεκριμένη τροπολογία. Τροπολογία 8 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κύριε Μπιάνκο. Πρόεδρε. Είμαστε σε μια φάση όπου στην Ευρώπη διαπιστώνουμε ένα πολύ έντονο φαινόμενο αστικοποίησης και το 1 τρίτο των πολιτών θα ζει πολύ σύντομα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η δική μου πρόταση προβλέπει στρατηγικές συγκεκριμένες με στόχο να προστατευτούν οι μικρές κοινότητες. Ως Επιτροπή των Περιφερειών εμείς πριν από λίγο καιρό μόλις εγκρίναμε μια ε, απόφαση, μια έκθεση η οποία θα φέρουν προς τους σπόρους στην προστασία των μικρών ε, κοινοτήτων. Ε, έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα μια προσοχή ιδιαίτερα στη διατηρήσει στρατηγική αυτή, την επικοινωνιακή κιόλας, που ε, αναγνωρίζει τη διαφορά μιας μικρής κοινότητας από ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Παρακαλώ του συναδέλφου τουλάχιστον τη πολιτική μου ομάδα να δώσουν κάποια ιδιαίτερη προσοχή και να δείξουν μερίμνα για τι μικρέ κοινότητε. Καλώ. Ψηφίζουμε τροπολογία αυτή. 8 ψήφι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι, υπέρ, είναι κατά, συγγνώμη, απορρίπτεται. Επομένω, πηγαίνουμε στην τροπολογία 9 ψήφι υπέρ. Κατά. Είναι υπέρ η περισσότερη, εκρίνεται η 9 και προχωρούμε στην 10 ψήφι υπέρ. Κατά. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 ψήφι υπέρ Ψηφίζουμε. Κατά. Λίγοι. Περισσότεροι είναι υπέρ. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Περισσότεροι είναι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Επαναλαμβάνω την ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ θα ψηφίσουμε. Yes or no. Yeah. And after this vote και θα διακόψουμε μετά από την ολοκλήρωση τη συγκεκριμένης ψηφοφορίας για να έχουμε τη συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Κατάινεν. Λοιπόν, κατά ήταν οι περισσότεροι, επομένω η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε. Θα συνεχίσουμε ε, αργότερα από την τροπολογία 14 και μετά. Και τώρα να καλωσορίσω το Γύρκι. Ε, Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά προσωπική γιατί έχω συνεργαστεί με τον Γύρκη στην ΕΣΠΟ, την πατρίδα μας, ε, την ε, και Σα στήριξα και όταν είχατε διατελέσει πρωθυπουργό της χώρας. Ε, σας ευχαριστώ που είστε εδώ για να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Μια συζήτηση που αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση λόγω της ε, μετάβασης θέλουμε οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης να είναι μια αρχή που θα καθοδηγήσει τις μελλοντικέ δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό είναι ένα σημαντικό ε, μήνυμα, το βλέπουμε και στη γνωμοδότηση κ. Μπραμβίτσιους που θα τη συζητήσουμε αργότερα, την ε, γνωμοδότηση Αρνόλντα Αμπραμαβίτσιους. 65% ή μάλλον να μην ε, μπω σε λεπτομέρειες Έχουμε 169 στόχους που λένε το, 100, 65% δεν μπορεί να το πετύχουμε αν δεν συμμετέχουν οι, ε, τα άλλα επίπεδα κάτω από το εθνικό ε, και αν δεν υπάρχει πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Η Επιτροπή των Περιφερειών ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ακούσει ποια είναι η δική σας άποψη για την μελλοντική εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ιδιώ τώρα δεν ξέρω αν έχετε λάβει το φυλάδιο της Φιλανδικής Προεδρίας. Αν όχι, σας το εγχειρίζω. Διότι κατά την επόμενη περίοδο έξι μηνών, κατά το επόμενο τα ακούσαμε και από ε, την Πρωθυπουργία της Φιλανδίας σήμερα, που προτεραιότητα είναι το κλίμα και η ε, στόχη βιώσιμης ανάπτυξη τη Φιλανδική Προεδρία. Πολλοί δήμοι, περιφέρειες η Νότια Φινλανδία, το Ελσίνκι, ενημερώθηκαν ότι είναι παριθμόν ένα στη καινοτομία και η Φινλανδία δεύτερη μετά την ε, προσδισμάς γείτονα χώρα Σουηδία. Η δεύτερη πατρίδα μας, η ΕΣΠΟ, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Φιλανδίας, ε, είναι ένας από τους πρωτοπόρους ε, στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, Είμαστε και σε ένα πρόγραμμα ε, ηγεσία ε, για τους στόχους αυτούς ε, υπήρχε και η διάσκεψη των πρωταθλητών των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο ΕΣΠΟ που παρευρεθήκαμε. Στηρίζουμε λοιπόν ενεργά αυτούς τους στόχους και τώρα σε ό,τι αφορά το θεματολόγιο, αυτό θα μας τα πει ο κύριος Κατάιν, που ποιος μπορεί να είναι εδώ μέχρι τις παρατέταρτο Θα ακούσουμε τη συζήτηση, την, ομιλία και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και θα ε, τα καταθέσουμε και επί χάρτου όλα αυτά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μάρκο, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που δίνετε αυτή τη δυνατότητα να συζητήσω μαζί σας για την βιωσιμότητα και τους ε, στόχους της. Πρέπει να ομολογήσω ότι κατά τη θητεία μου η Επιτροπή έχει αλλάξει μερικά τις μεθόδους εργασίας της και μία από τις αλλαγές ήταν να αυξήσουμε και να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας με τις πόλεις και τις περιφέρειες. Γιατί αντιληφθήκαμε ότι πολλοί από τους στόχους μας εξαρτώνται από την ε, ενεργό συμμετοχή και τις καινοτομίες που εισάγουν οι πόλεις, οι δήμαρχοι, οι περιφέρειες. Γι' αυτό δημιουργήσαμε διάφορες ε, συνεργατικές πλατφόρμες μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και Πόλεων. Για παράδειγμα, η κυκλική οικονομία. Οι πόλεις είναι στην πρώτη γραμμή. Δημιουργούν ε, νέους τρόπους ε, αντιμετώπισης των αποβλήτων και νέε διαδικασίες δημοσίων προμηθειών για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό πάντα χαίρομαι ιδιαίτερα όταν συμμετέχω στις εκδηλώσεις, στις συνεδριάσεις σας. Γιατί θεωρώ ότι η Επιτροπή των Περιφερειών, οι πόλεις μας, είναι κύριος εταίρος μας για να εφαρμόσουμε την πολιτική μας, τις καινοτομίες μας. Αν δεν υπάρχει αυτή η στενή σύνδεση, δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Δύο λόγια τώρα για την πολιτική μας για τους στόχους της βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Κοιτάξτε, είναι στο γονιδίωμά μας ε, η βιωσιμότητα. Αν δείτε τις πολιτικές μας, για παράδειγμα, το διαπιστώσετε, η βιωσιμότητα είναι τμήμα του γονιδιώματός μας. Θέλουμε να συνεργαστούμε και να εργαστούμε με δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα οι στόχοι αυτοί να είναι κεντρικό στοιχείο όλων μας των πολιτικών και των προτεραιοτήτων της Επιτροπής. Και το δεύτερο στοιχείο της πολιτικής μας είναι αυτό το έγγραφο προβληματισμού, στο οποίο θα επανέλθω. Πρώτα απ' όλα, πώς θα ενταχθούν σε όλες μας τις πολιτικές. Η Επιτροπή μας έχει βάλει την ε, βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις οριζόντες πολιτικές, αλλά και σε κλαδικές πολιτικές και πρωτοβουλίες. Ορισμένα παραδείγματα αυτό των κλαδικών πολιτικών. Η κυκλική οικονομία είναι για παράδειγμα παράδειγμα. Κάνουμε βήματα λοιπόν για να αλλάξουν ε, οι τρόποι παραγωγής και κατανάλωσης. Εστιάζουμε περισσότερο στο σχεδιασμό των προϊόντων, τη διαχείριση των αποβλήτων και την αύξηση της ε, Τα πλαστικά τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έτσι θα προστατεύσουμε το περιβάλλον και θα προωθήσουμε και την ανάπτυξη και την καινοτομία. Και η νέα ε, πολιτική μας για την βιοοικονομία θα βοηθήσει την καλύτερη χρήση των ανανεωσίμων. Επίσης, βιώσιμη χρηματοδότηση. Θεωρώ ότι οι πρωτοβουλίε για το στόχο αυτό της βιώσιμης ε, χρηματοδότησης ίσως είναι η σημαντικότερη μεμονωμένη πρωτοβουλία για να αλλάξει ο κόσμος. Και το πρόγραμμα επενδύσεων για την Ευρώπη ανέπτυξε τις ε, επενδύσεις μας για τις ανανεώσιμες, την κυκλική οικονομία, την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τώρα, αυτό το έγγραφο προβληματισμού για μια βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030. Είναι το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο φέτος μαζί με τον Αντιπρόεδρο Φρανς Τίμερμανς. Το έγγραφο είναι τμήμα της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Στόχος του είναι να εμπνεύσει τη συζήτηση για τις πολιτικές προτεραιότητες μετά το 2019 περιέχει διάφορες αναλυτικέ λύσεις με διάφορες ιδέες για να προωθήσουμε τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον εισηγητή Αρμάντα Αμπραμιβίτσιου και όλα τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ για το σχέδιο γνωμοδότησης και για το ότι είχαμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την έκθεσή σας. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Αυτό ακριβώς θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να προωθήσει την συζήτηση, να συλλέξουμε σωστές ιδέες για να αναμορφώσουμε τις πολιτικές μας για την επόμενη θητεία. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη σκληρή εργασία σας. Και για το θέμα αυτό. Τέλος. Η τοπική εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, η, το θεματολόγιο του 2030 και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ε, είναι ακριβώς το πρόγραμμα που πρέπει να ε, εφαρμόσουμε όλοι η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας, ο πανεπιστημιακός τομέας αλλά και οι πολίτες γενικά. Το θεματολόγιο του 2030 υπογραμμίζει ότι το να υιοθετήσουν τα κράτη αυτό το πρόγραμμα έχει τεράστια σημασία για την επιτεύξη βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δημόσιες οι αρχές, οι κρατικές αρχές, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό μπορούν να διδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Και αυτό είναι το πεδίο δράση του δικό σας. Και επίσης όπως επισημαίνεται άλλωστε και στο σχέδιο γνώματο της Επιτροπής 65% από τους 169 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη μπορούν να αναπτυχθούν, πρέπει να αναπτυχθούν σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό για να επιτευθούν οι στόχοι τους σε υποεθνικό λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο πρέπει να αναπτυχθεί και να γίνει πραγματικότητα η βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει και συμμετοχή, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση. Σημαίνει ότι τον κύριο ρόλο θα έχουν να τον διαδραματίσουν οι τοπικές και περιφερειακές, υπό, ε, οι αρχές κάτω από το επίπεδο της εθνικής διακυβέρνησης. Και θα αναφερθώ και στο παράδειγμα που έδωσε ο πρόεδρο. Η περιφέρεια τη Ούζημα στην Νότια Φιλανδία έχει προβληθεί ω υπόδειγμα. Και γιατί το λέω αυτό, όχι γιατί το είπε ο πρόεδρο, όχι γιατί είμαι Φιλανδό. Αλλά γιατί την καινοτομία την κοινή την προβάλλει η περιφέρεια. Μια η αδίποτε καινοτομία έλαβε χώρα σε μια η αδίποτε συγκεκριμένη περιφέρεια και γι' αυτό είναι καλό να υπάρχει αυτή ε, ο συναγωνισμός μεταξύ των περιφερειών για τους ε, ε, στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χωρί αυτόν τον συναγωνισμό, χωρί αυτή την άμυλα, δεν μπορούμε να έχουμε την επίτευξη τη πρόοδου, βέβαια και των στόχων. Το λάχτη επίση, ίσως να ξέρετε ότι έχει επιλογή, επιλογή ως πόλη πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης, όχι λόγω των ε, στόχων αυτών ε, συγκεκριμένα, αλλά γιατί είναι μια πόλη ότι, ε, η οποία έχει μπορέσει να κάνει καθαρισμό των λίμνιων υδάτων. Δηλαδή, όποιος περπατάει στην όφτα της λίμνης μπορεί να βάλει στο χέρι του νερό και να το πιει. Χρησιμοποιεί επίσης μόνο ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ενέργειας και πολλά άλλα πράγματα. Αν δεν είχαν γίνει αυτέ οι προσπάθειε σε τοπικό επίπεδο, κάποιε από τι καινοτομίε που δημιουργήθηκαν και κάποια επιχειρηματικά μοντέλα δεν θα υπήρχαν. Και έτσι δεν θα υπήρχε και η ανάπτυξη που στηρίζεται σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο. Σε αυτό θέλω να τονίσω και να εξαρώ τη σημασία τη ε, τοπική ε, και περιφερειακή διακυβέρνηση για την επίτευξη των στόχων. Uh, Καλώ ευχαριστώ πολύ τονίσατε στην ομιλία σας τι σημαίνει η δική μας η διάσταση, πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε. Σύντομες παρεμβάσεις τώρα από τις πολιτικές ομάδες με πρώτο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριος Άμπραμοβίτσιους ο συζητητής, έχει το λόγο. Σα υπενθυμίζω βέβαια πως έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο για να προλάβει και ο Αντιπρόεδρος να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάκουλα την Πρόεδρε, κύριε είναι εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, θέλω να σας και τη πολιτική του ομάδα. Εδώ θέλω να σα καλωσορίσω στην Επιτροπή των Περιφερειών. Σα ευχαριστώ για την τοποθέτησή σα, για τα θέματα που αφορούν εμένα ιδιαίτερα ω εισηγητή για του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη πολύ ε, επίπεδη διακυβέρνησης και να πω ότι είναι πολλές οι προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν οι πόλεις, οι περιφέρειες για να μπορέσουν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης. Σήμερα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε αυτές ακριβώς τις προκλήσεις και θα ήθελα ξεκινώντα να επισημάνω πως χρειάζεται να υπάρξει, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια βάση κατάλληλη για την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να προβάλλει ένα συγκεκριμένο σχέδιο με τον τίτλο Σενάριο 1 όπως το έχουμε ήδη περιγράψει με μια στρατηγική ευρεία κάλυψη που θα ορίσει συγκεκριμένου στόχους και ορόσημα που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο 2030. Επίσης έτσι θα έχουμε και το πλεονέκτημα να ξεπερνούμε τους κύκλους της πολιτικής εναλλαγής και να προχωρούμε όλοι ταυτόχρονα με τους στόχους αυτούς που μπορούν να επιτρέψουν στην Ευρώπη το 2030 να υλοποιήσει τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που έπεται. Επίσης χρειάζεται η ε, ενεργό συμμετοχή των ε, αρχών σε επίπεδο κάτω από την εθνική διακυβέρνηση στην επίτευξη των στόχων. Επίσης θα πρέπει η στρατηγική αυτή να, επιτύ... να στηριχθεί σε ουσιαστικές επενδύσεις που μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές και διαφορά μέσα. Η πολιτική συνοχή είναι πιο σημαντική, ε, το πιο σημαντικό μέτρο για την εισαγωγή επενδύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση με στόχο την επίτευξη των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Άλλα μέτρα όμω υπάρχουν και μπορούν και αυτά να ε, ε, αξιοποιηθούν με την ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης όπως σε παραδείγμα την κατευθύνηση γραμμές για την καλύτερη νομοθεσία. Και θα ήθελα να δώσω παράδειγμα από το Δήμο μου, από το Ζαγασέι της Λιθουανίας, μικρό Δήμο, που όμως μαζί με άλλους δήμους της Λιθουανίας έχει μπορέσει να εισαγάγει και να εφαρμόσει ένα συνολικό πρόγραμμα για την ανακαίνιση των ε, οικίσκων ε, του Σοβιετικού συστήματος, του παλαιού συστήματος, έτσι ώστε και να καταστούν πιο οικονομικοί ε, ενεργειακά, οικονομική ενεργειακά αυτή η κίσκη, που βεβαίως το χρειαζόμαστε για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και που το χρειάζεται και ο πιο φτωχό πολίτης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ΕΣΠΟ επίσης, ένας άλλος δήμος, έχει ορίσει σαν στόχο να προχωρήσει στην υλοποίηση των ε, δεσμεύσεων και των στόχων ε, πέντε χρόνια νωρίτερα από ό,τι έχει προβλεφθεί. Αυτό το κάνουν και άλλες ε, κοινότητες και δήμοι στην περιφέρεια μας. Ρωτώ λοιπόν πώς βλέπετε αυτή την εικόνα και πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε κατόπιν της εφαρμογής του, νέας στρατηγικής, του νέου στρατηγικού θεματολογίου από την Προσεχή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για να ξαναπεράσω στη διαδικασία της υλοποίησης αυτής της στρατηγικής, αναφερόμενος και σε κάποια άλλα στοιχεία που μπορεί να συμβάλλουν στην επιτυχία της, ε, όπως λέγαμε και νωρίτερα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη δουλειά μας σε επίπεδο, να συνεχίσει τη δουλειά της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια στο δικό της επίπεδο. Η μορφή της συνεργασίας που θα έχουμε έστω και διαφοροποιημένη θα πρέπει να είναι υπαρκτή, θα πρέπει να είναι ουσιαστική και σε μια πλατφόρμα με συμβολή πολλών παραγόντων και φορέων νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. PES με τον κύριο Κούρτ. Τρία λεπτά. Πρόεδρε, εξωτιμοί κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ από την ομάδα μου να πω δύο λόγια. Από την εμπειρία που έχουμε για την, από την εφαρμογή ενός μοντέλου με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Ξεκινώ καταρχά με τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο το σενάριο υπαριθμών 1 είναι αυτό το οποίο μπορεί πράγματι να μα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, ένα βιώσιμο μέλλον και δίνει τον κατάλληλο προσανατολισμό μια στρατηγική η οποία δεν ε, ισοδυναμεί με το άθροισμα διαφορετικών πολιτικών. Δηλαδή θα λέμε «Α, κάνουμε αυτό για το περιβάλλον, άντε να κάνουμε και κάτι για την οικονομία ή τούμπαλιν», αλλά του αντίον ε, μια στρατηγική, μια πολιτική που θα είναι μια συνεπής πολιτική, μια ολοκληρωμένη πολιτική και που θα μα επιτρέψει να έχουμε ε, ένα σύνολο αποτελεσματικό. Επίση, πολιτική για την αηφορία δεν είναι απλώ μια πολιτική αηφορία. είναι μια πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει και χαρακτήρα αηφορία. Άρα δεν έχουμε την αηφορία σε ένα χωριστό ε, τμήμα, αλλά ενσωματώνεται αυτή μέσα σε κάθε άλλη πολιτική και η διάσταση που μα απασχολεί είναι η μεταμόρφωση του οικονομικού συστήματος και του τρόπου διαβίωσης κατά τρόπο ώστε να καταστεί αηφόρο βιώσιμο. Έχουμε μια εμπειρία 300 ετών με την δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας και τη οικονομική ανάπτυξη που όμω πολλέ φορέ δεν συνοδευόταν από μια βιώσιμη πολιτική και άρα πρέπει να βρούμε μια νέα πολιτική και άρα ορίζουμε στόχου. δεν στηριζόμαστε μόνο στου τεχνοκράτε και μόνο στα ει δυνάμεις της αγοράς, προχωρούμε σε μια μεταμόρφωση η οποία είναι απαραίτητη και η οποία θα έχει χαρακτηριστικά αηφορία. και πρέπει να είμαστε εμεί εκεί παρόντε. είναι μεγάλη η πρόκληση. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα θέλαμε. Ε, πιέζει ο χρόνος, το 2030 είναι αύριο και γι' αυτό πρέπει να ε, ανοίξουμε το βήμα. Η πολιτική λοιπόν ε, αυτή η οικονομική δεν είναι παρά ένα μόνο κομμάτι, ένα στατικό στοιχείο, ένα τουβλάκι μέσα στην πολιτική τη ε, βιώσιμης ανάπτυξη και δεν, μπορεί να λησμονηθούν, δεν μπορούν να λησμονηθούν τα υπόλοιπα τουβλάκια, τα υπόλοιπα στοιχεία όπω η πολιτική για την προσέγγιση του περιβάλλοντος ή η κοινωνική πολιτική. Αν αυτά λησμονηθούν δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Άλλη μια παρατήρηση που έχει να κάνει με την διακυβέρνηση, με τη λογοδοσία, με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Θα ήθελα να δώσω ένα θετικό παράδειγμα το θεματολόγιο για τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωση που μπορεί να αποτελέσει, που οφείλει να αποτελέσει έναν προσανατολισμό για τους τρόπους συνεργασίας και ιδιαίτερως ευχαριστώ για τις δυνατότητε που έχουν τα ε, οι δήμοι, κοινότητες να μιλήσουν, να συνομιλήσουν, να καταστούν ε, συνομιλητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2020 του χρόνου δηλαδή θα γίνει μια μεγάλη διάσκεψη των ε, πόλεων. Ε, δήμων και Κοινότητων, δηλαδή στην ιδιαίτερη μου πατρίδα του Μανχάιμ και θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε νομίζω τι προτάσει για τη μεταμόρφωση και το χαρακτηριστικό της πολυεπίπεδης διακυβέρνηση που θέλουμε να έχει αυτή. Ευχαριστούμε από την Άλντε η Renew Europe όπως λέγεται πλέον. The Βερφαλή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο τη Κομισιόν για την παρουσίαση. Το θέμα μα είναι ο εντοπισμό των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη ε, στην Ένωση. Πολύ σημαντικό θέμα. Οι τοπικέ περιφερειακέ αρχέ αναπτύσσουν και θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν σχέδια, να ξεχρονίζουν υποδομέ, εργάζονται και θα εργάζονται σε συνεργασία με τον πολίτη για την επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Ήδη βιώνουμε τι αρνητικέ συνέπειε τη αλλαγή του κλίματο. Φυσικά φαινόμενα ακραία πιέζουν τι δυνατότητε που έχουμε να εγγυηθούμε τις δημόσιες υπηρεσίες. Η γνωμοδότηση του συναδέλφου ε, αναφέρει και τα σενάρια ε, που έχει προτείνει η Κομισιόν, ένα από τα οποία είναι και το μόνο βιώσιμο για να εγγυηθούμε την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στην Ένωση. Να τονίσω τα μέτρα ιδίω για την ε, ιδιοποίηση της κυκλικής οικονομίας ό,τι αφορά το δεύτερο ισοζύγιο άνθρακα. Θα πρέπει να είναι κλειδί της βιομηχανικής στρατηγικής η βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων και η Ζανέτ Μπαλιέ την κυκλική οικονομία τη βάζει στο επίκεντρο της γνωμοδότησής της σε ό,τι αφορά την εδαφική προσέγγιση. Η κυκλική οικονομία είναι σημαντική, ε, σημαντική προτεραιότητα και ευκαιρία για τις ε, τοπικές αρχές. Δημιουργούνται έτσι ε, θέσεις εργασίας ε, που δεν θα μπορούν να μετεγκατασταθούν. Θα έχουμε νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις. Θα πρέπει να δούμε διαφορετικά την καινοτομία, να στοχαστούμε νέες υπηρεσίες, νέα αγαθά, να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και θα πρέπει η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη διαβίου μάθηση να είναι εγγυημένη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις τεχνολογίες των πληροφοριών που θα έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Βελτιστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, παράγουμε. Θα χρειαστούν μαζικές επενδύσεις για να προσαρμόσουμε τα δίκτυα στις ανάγκες της κυκλικής οικονομίας και αυτό πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο. Ο εντοπισμό των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη θα απαιτήσει πιο στενή συνεργασία μεταξύ κοινών πολιτών, βιομηχανία, ΟΤΑ, σχολείων, πανεπιστημίων για να να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να είμαστε όμω και στη σωστή κατεύθυνση θα πρέπει τα χρήματα της Ένωση να τα αξιοποιούμε μόνο όταν αυτά προωθούν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι στόχοι ουσιαστικά είναι ε, μια βιώσιμη ε, αναπτυξιακή στρατηγική και πρέπει να συνεχίσουμε να τους εφαρμόζουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μπορέλ Πόρτα. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία αυτή και θέλω να σας πω ότι γίνεται στη Βαρκελόνη. Η Καταλωνία γενικά ε, είναι προσιλωμένη στους στόχους ε, του 2030 και στο διεθνές επίπεδο και στο δίκτυο για την περιφερειακή διακυβέρνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμμετείχαμε ενεργά και στον ορισμό των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο εσωτερικό ο στόχο μας είναι όλοι οι φορείς να συμμετέχουν, που είναι βασική άλλωστε αρχή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν φορεί οι οποίοι συμμετέχουν από την αρχή όπω το νομοδοτικό Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Καταλονίας που έχει κάνει και μια έκθεση για την μεταρρύθμιση Καταλωνίας και τη βελτίωση του κόσμου, στόχοι και θεματολόγιο το 2030. Πριν δύο χρόνια η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα σχέδιο εφαρμογή αυτών των στόχων με όλα τα καταλανικά υπουργεία. Τον Ιούλιο θα εγκριθεί και θα μιλάμε για την πραγμάτωση των 17 στόχων με 80 ε, στόχους, ε, μάλλον 800, 800 project συγκεκριμένα. Επίσης δεσμευόμαστε ως κυβέρνηση για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης κάθε δύο χρόνια θα εξηγεί το τι έχει πετύχει και θα υπάρχουν επίσης περιοδικές επαφές ε, με τα περιφερειακά υπουργεία, στα οποία επίσης θα παρουσιάσουν τι έχει γίνει μέχρι στιγμής στο επίπεδο της Καταλωνίας. Η Καταλωνική κυβέρνηση επίσης ε, καταρτίζει και μια εθνική συμφωνία για να έχουμε μια ε, σύμπραξη δημόσιο-δικοτικού τομέα σε ειδικά θέματα που άπτονται των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω ολοκληρώνοντα να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Περιφερειών που θέλει να ενισχύσει το ρόλο μα για την ε, βελτίωση του θεματολογίου. Ευχαριστώ το ΕΣΥΑ. Ο κύριος Ότιλ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είναι ουσιώδες συζήτηση αυτή να υπογραμμίσουμε επαρκώς ότι η στρατηγική το 2030 στοχεύει στην αντιμετώπιση των απειλών που έχουν να κάνουν με την παγκοσμιοποίηση. Η στρατηγική αυτή έχει παγκόσμια διάσταση και φιλόδοξους, πολύ φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και για την οικονομία μας. Ο πρόεδρος Μάρκου Μάρκουλα τόνισε ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης περιέχουν 169 ε, μέτρα εκ των οποίων το 65% πρέπει να υλοποιηθούν με τη συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Άρα είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο μα. Πρέπει να το σημειώσουμε. Πρέπει ακριβώ να εμπλακούν οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ στην εφαρμογή των στόχων αυτών γιατί είναι αυτοί οι φορείς, οι αρχές που είναι πιο κοντά στους πολίτες πολύ εύκολα λοιπόν, πολύ ευκολότερα μπορούν να εντοπίσουν τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί η επιρροή τους στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών. Η στρατηγική μας για το 2030 συνδυάζεται με την πολιτική συνοχής που σύμφωνα με τις συνθήκες πρέπει να στοχεύει στην εξίσωση του επίπεδου ευημερία των διαφόρων περιφερειών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει λοιπόν να παίξουν ε, μεγάλο ρόλο στην πολιτική συνεχής, συνοχή και να συνεχίσουν και στο μέλλον. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απειλή για ε, τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. Από σήμερα πρέπει να δράσουμε, από σήμερα πρέπει να εφαρμόσουμε τις πολιτικές αυτές, αλλά με ιδιαίτερα σόφρονα τρόπο για να μην παρεμποδίσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης των μελλοντικών γενεών. Έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχει συλλογικά η ευρωπαϊκή κοινωνία. Για παράδειγμα, οι μακροπεριφερειακέ στρατηγικέ. Όλε αυτέ οι νέε δυνατότητε πρέπει να ενισχυθούν και να εφαρμοστούν πολύ περισσότερο. Κάιζερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η βιωσιμότητα χρειάζεται συγκεκριμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα, στο Κέρνταν, στην Καρινθία, στην Αυστρία, λέμε ότι οι πόροι μα πρέπει να χρησιμοποιούν τόσο πολύ ώστε τα παιδιά μα, τα εγγόνια μα να έχουν και στο μέλλον ένα υγιές περιβάλλον. Για να το κάνουμε αυτό, στην Καρινθία θα λάβουμε δημοσιονομικές και πολιτικές αποφάσεις που σχετίζονται με και συμμορφούνται με τους στόχους ε, του ΟΗΕ. Βεβαίως η οικονομία. Και ο κάθε πολίτης πρέπει να έχουν υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλευόμεθα με ληστρικό τρόπο τους πόρους μας. Πρέπει να γίνουμε από dreamers and doers, δηλαδή από αυτούς που ονειρεύονται σε ανθρώπους της δράσης. Τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να μην έχουμε ε, άσωτη ποσοτική ανάπτυξη, αλλά αντίθετα με στόχο τη βιωσιμότητα να αντιμετωπίσουμε τον νέο φιλελευθερισμό. Ιδιαίτερα όλες οι περιφέρειες και τα κράτη χρειάζεται να συμμετάσχουν. Και τώρα η συγγήτρια Σύρπα Χέρτελ. Είναι επίσης ε, συγγήτρια και για την άλλη γνωμοδότησή μας που θα συζητήσουμε τον Οκτώβριο για τους βιώσιμους στόχους. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Επίτροπε κύριε Κατάινεν. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα να συζητήσουμε την ε, υλοποίηση των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαι η συγγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της έκθεσης για το κλίμα και την ενέργεια ως πτυχές της ε, επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030. Ταυτόχρονα είμαι και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΕΣΠΟ που επιλέγει πριν από την ε, καταρρεπτική προθεσμία του 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα μάλιστα, να έχει φτάσει στους στόχους. Θέλω λοιπόν εκ μέρου τη Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και εκ μέρου της ε, ιδιαιτερής μου πατρίδας τη ΕΣΠΟ να διατυπώσω τα ερωτήματα. Χρειάζεται, κύριε Επιτροπέ, μια σαφή ευρωπαϊκή στρατηγική για του στόχου τη χιλιετία με μια ολιστική προσέγγιση ω προ την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα Δεύτερον, οι πόλεις και οι περιφέρειες έχουν ε, τη δυνατότητα να υλοποιήσουν μέχρι και 60% των στόχων, έχοντας από την άλλη το 30% της χρηματοδότησης και τον πέμπτο των δημοσίων επενδύσεων των σχετικών με τους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, δεν πρέπει να συνεργάζεται το, η κεντρική κυβέρνηση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης, εμείς υλοποιούμε, μετατρέπουμε σε πραγματικότητα στο, στο Δήμο μας, στην κοινότητά μας αυτούς τους στόχους και άρα χρειάζεται, ε, χρειαζόμαστε εργαλεία που μας επιτρέπουν την αξιολόγηση της πρόοδου και ταυτόχρονα χρειάζεται η κλιματική αλλαγή να βρει αντανάκλαση και στη δημόσια χρηματοδότηση, στην κρατική χρηματοδότηση. Είναι όλα αυτά στόχοι που πρέπει να προβάλλουμε. Επίσης θα γίνει στο ΕΣΠΟ στις 8 ε, Ιουλίου ένα σεμινάριο για την ε, συζήτηση συγκεκριμένων δράσεων προς την επίτευξη των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης για να έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικές στη χρήση ενέργειας με περισσότερη βιοπικιλότητα ε, πόλης, κομμαπόλης και χωριά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, σας περιμένουμε στο ΕΣΠΟ στις 8 Ιουλίου σε μια συζήτηση που πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ Σύρπα και τώρα παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο Γιούρκη Κάτα να λάβει το λόγο για να δώσει απαντήσεις στα σχόλια που ακούστηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις και μου πέφτει εύκολο να συμφωνήσω με τις ιδέες ε, που ακούστηκαν. Εγώ θα ήθελα ωστόσο να σταθώ σε πέντε σημεία. Αυτά τα οποία αν ήμουν εγώ ο, να, αρμόδιος για τη λήψη των αποφάσεων μόνος μου στην Ευρώπη θα εστίαζα. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στην εκπαίδευση που είναι ο μόνος και ουσιαστικός τρόπος εξασφάλισης κοινωνικής ε, δικαιοσύνης, βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης των πολιτών, και ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Είναι ο καλύτερο και πιο σοβαρός τρόπος να πείσουμε τον πολίτη να κάνει καλύτερες αλλά και πιο συνειδητές επιλογές και να εγκαταλείψει αυτά που θα μπορούσε ενδεχομένω να κάνει λάθος ε, σε θέματα περιβάλλοντος. Δεύτερον, θα ενίσχυα τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, ώστε να συνδυαστεί με τους αντίστοιχους των περιφερειών μας, προϋπολογισμούς για την έρευνα, και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα των κονδυλίων που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές οι περιφέρειες και οι Δήμοι και γι' αυτό το ορίζον Ευρώπη έχει τόσο σημασία να το στηρίξετε και εσείς. Εκεί προτείνουμε την αύξηση της ε, χρηματοδότησης για την έρευνα. Ένα ζήτημα και μια επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα για την Ευρώπη. Τρίτον, θα ήθελα περισσότερο να εστίαζα και ελπίζω να το πράξει ο επόμενο ε, επίτροπο, στην κυκλική οικονομία που έχει ιδιαίτερα ε, ε, για την οποία έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο οι δήμοι, οι κοινότητε. Ξέρετε πολύ καλά και από εσά, από τι δικέ σα δημοτικέ επιχειρήσει, ότι πρέπει και εσεί να επιδείξετε ή να ακολουθήσετε τι βέλτιστε πρακτικέ, αλλάζοντα και κάποιε διατάξει ενδεχομένω, όπω μπορεί να γίνει για να προαχθεί η κυκλική οικονομία στο δικό σα επίπεδο ήδη. Τέταρτον, και αυτό ίσως να είναι και η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη, η υποβάθμιση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Δυστυχώς, σήμερα η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι κάποιοι από τους πολιτικούς ταγούς θεωρούν πως η φιλελεύθερη δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι μια αντίληψη του παρελθόντος, παροχημένη. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό όμως διότι δεν μπορεί να υπάρξει ε, πρόοδο στην Ευρώπη, δεν μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα ε, και ανάπτυξη εάν δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δημοκρατία και ελευθερίες. Και σε αυτό χρειαζόμαστε πάλι την ε, προστασία αυτών των θεμελιωδών αξιών και από τους δήμους και τις κοινότητες. Και εν τέλει θα ήθελα να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Σε όρους τεχνολογικούς είναι σημαντικό να επενδύσουμε περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Το ίδιο όμω ισχύει και ε, για λόγους ε, προσφοράς ε, δημοσίων υπηρεσιών. Γιατί αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ε, ποιότητα τη γνώση αλλά και των δεδομένων που έχουμε στη θέση μα, μπορούμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρουμε στον πολίτη και την αποδοτικότητα αυτή τη ε, παροχή υπηρεσία. Και αυτή είναι μία πτυχή τη τεχνητή ε, νοημοσύνη και υπάρχει και η άλλη πτυχή τη τεχνητή νοημοσύνη που λέει και ανησυχεί ότι μπορεί να έχει χαρακτήρα διατάραξης της οικονομικής, ανατροπής λέει, της οικονομικής ε, κατάστασης η τεχνητή νοημοσύνη και μας λέει ότι θα χαθούν ενδεχομένως πολλές θέσεις εργασίας. Αυτούς δεν μπορούμε να τους λησμονήσουμε. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε αυτούς ε, των οποίων το επάγγελμα θα εξαφανιστεί λόγω ίσως της ε, ε, τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορούμε να λησμονήσουμε αυτούς των οποίων το επάγγελμα θα εξαφανιστεί γιατί δεν έχει γίνει πιο σύγχρονη η ε, εκπαίδευσή μας που, που τους προσφέρουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρουν μια θέση εργασίας καινούρια, να μπορέσουν να ξεφύγουν από το πρόβλημα της ανεργίας πριν να είναι πολύ αργά. Και έτσι κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσω μέσα σας και ελπίζω βέβαια να παραμείνουμε σε στενή επαφή από εδώ και στο εξή σε ό,τι αφορά τα πέντε σημεία που αναφέρατε. Πρέπει να σας πω ότι για την παιδεία ιδίω έχουμε πολλές γνωμοδοτήσεις, το στηρίζουμε το θέμα αυτό. Ο Κριστόφερ είναι ένας από τους ε, συγητές μας. Ε, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ε, πάνω στο θέμα αυτό για να καταλήξουμε και να φτάσουμε εκεί που είπατε εσεί Το δεύτερο, η κυκλική οικονομία, πράγματι και το κράτος δικαίου είναι σημαντικό κομμάτι των γνωμοδοτήσεων με τον για τη πολιτική βούληση, βέβαια και ψηφιοποίηση που επίση αναφέρατε είμαι εισηγητής για την ε, ψηφιακή Ευρώπη και η συνάδελφος από τη Φινλανδία ε, επί Φινλανδικής Προεδρίας ε, θα αναλάβει το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλά και ελπίζουμε όλα αυτά να τα συνδέσουμε και με τους στόχους που Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Είχα πει πριν ότι όποιοι θέλετε να συνεισφέρετε μπορείτε είτε τώρα να το πράξετε είτε όταν θα έχουμε τη συζήτηση για την γνωμοδότηση του κυρίου Αρνόλντας Αμπραμιβίτσιους. Επειδή το θέμα είναι το ίδιο λίγο πολύ. Θέλει κανείς τώρα το λόγο ή όταν θα έρθει η ώρα της έκθεσης του κυρίου Αμπραμαβίτσιου. Σας προχωρήσουμε έτσι. Και να επανέλθουμε τώρα στην ψηφοφορία του σχεδίου, επί του σχεδίου ψήφισματος. Ήμασταν στην τροπολογία 14, τη θέτω σε ψηφοφορία Hans Christian Jessens και λοιποί. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Ωραία, ψήφι υπέρ. Πολύ 14. Κατά τώρα. Είναι κατά οι περισσότεροι, άρα απορρίπτεται η τροπολογία 14. Τροπολογία 15. Οι σοσιαλιστές θέλουν χωριστή ε, ψηφοφορία, σε τμήματα δηλαδή. Μιλάν, Μιλάνα, παρακαλώ εσείς να μας το παρουσιάσετε. Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια τροπολογία που έχει να κάνει με την χωριστή ψηφοφορία. Εδώ έχουμε μια. Έχουμε ζητήσει δηλαδή τη χωριστή ψηφοφορία σε τμήματα και έχουμε μια δυσκολία και θα ήθελα να γίνει μια διευκρίνηση στο δεύτερο τμήμα αυτή τη τροπολογία, ώστε να γίνει, να γίνει πιο σαφέ, πιο απλό κιόλα, πιο ισχνό. Και εφόσον συμβαίνει αυτό, μπορούμε να ανακαλέσουμε την, σε τμήματα ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν λέμε ότι θα θέλαμε ένα σύστημα ε, νομοθετικό στην Ευρώπη με βάση τους κανόνες που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη ε, για τους μισθούς και τους εργαζομένους. Αυτό θα αντικαθιστούσε το δεύτερο τμήμα. Και αυτό γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα έγγραφο το οποίο ε, αποτελεί την εισαγωγή του θέματος στο δημόσιο διάλογο. Στέλνουμε, στέλνουμε ένα έναυσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε μια αναλυτική επεξήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είναι μόνο μια αρχή, ένα έναυσμα και μια, ε, ένας προσανατολισμός για την Επιτροπή και νομίζω ότι αυτό αρκεί. Ευχαριστώ ο κύριος Ρίου. Η σοσιαλιστική ομάδα υποστηρίζει τη θέση αυτή του συναδέλφου, του κύριου Μιλάνα. Ω προ την ε, τροπολογία του. Καλώ. Άρα γίνεται σε τμήματα ψηφοφορία. Λοιπόν, πρώτο τμήμα σημειώνει και τα λοιπά μέχρι την, τις οικογένειές τους. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την πρώτη αυτή, το πρώτο σκέλος της τροπολογίας αυτής. We can close. ψηφοφορίας. Είναι υπερπερισσότεροι. περισσότεροι. Επομένω εγκρίνεται το πρώτο τμήμα και προχωρούμε στο δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Α, όχι, κύριο Μπορ. Αν κατάλαβα καλά, Πρόεδρε, είναι ότι το δεύτερο τμήμα είναι αντικείμενο προφορικού συμβιβασμού. Υποθέτω αυτό ψηφίζουμε τώρα, το κείμενο. Πρόεδρος, ναι, βεβαίως, προφορικός συμβιβασμός που όμως δυστυχώς δεν έχουμε επί της οθόνης, αλλά Νομίζω είναι γνωστό το κείμενο. Εντάξει, επομένως ψηφίζουμε το συμβιβαστικό κείμενο. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Υπέρ είναι η περισσότερη, επομένως ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Περισσότερο υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Ψήφι υπέρ. Κατά. Περισσότερο υπέρ. Τροπολογία 20. Συγγνώμη, διορθώνει. Ο πρόεδρος, τροπολογία 19. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ουδής εγκρίνεται. Τροπολογία 20 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ε, η τροπολογία απορρίπτεται. 21 ψήφι υπέρ. Κατά. Πλειοψηφία υπέρ. Επομένω εγκρίνεται. Τροπολογία 22 ψήφι υπέρ. Κατά. Λίγοι. κατά υπέρ, στο υπέρ εγκρίνεται τροπολογία 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Οι περισσότεροι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Περισσότεροι είναι υπέρ. Εγκρίνεται η 24. Τροπολογία 25. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 27 ψήφι υπέρ. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 ψήφι υπέρ. Κατά. Είπε στον κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 ψήφι υπέρ. Κατά περισσότερο υπέρ εγκρίνεται. 30. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 31. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται γιατί περισσότερο ήταν υπέρ. Τροπολογία 32. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 33 ψήφι υπέρ. Ναι, ευχαριστώ. Κατά. Ουδής εγκρίνεται. Τροπολία 34 ψήφι υπέρ. Κατά. Ουδής εγκρίνεται. Τροπολία 35 ψήφι υπέρ. Κατά. Ουδής εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Ουδής. Εγκρίνεται. 37. Ψήφι υπέρ. Κατά. Λίγοι. Περισσότεροι είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Προφορικό συμβιβασμός ε, για τις τροπολογίες 38 και 39 επί της οθόνης. Μπορούμε να ψηφίσουμε παρακαλώ. Αν εγκριθεί αυτός ο προφορικός συμβασμός οι 38, οι 31 και το πρώτο με 40 καταπίπτουν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Είναι υπέρ η πλειοψηφία. Επομένω εγκρίνεται και αυτό σημαίνει ότι 38, 31 και πρώτο στο τμήμα τη 40 καταπίπτουν. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 40 από τη λέξη ταυτόχρονα και μετά ψηφίζουμε ψήφι υπέρ κατά είναι κατά οι περισσότεροι συνάδελφοι απορρίπτεται τροπολογία 41 ψήφι υπέρ κατά υπέρ οι περισσότεροι εγκρίνεται 42 ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται 43 ψήφι υπέρ ευχαριστώ κατά ουδής εγκρίνεται και τώρα η τροπολία 44 ψήφι υπέρ κατά εγκρίνεται γιατί κανείς δεν ήταν κατά το σύνολο του ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί. Ψήφι υπέρ, κατά. Επτά, οκτώ, αποχές, μία. Ωραία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία και συγχαίρουμε αυτούς και αλλήλους. Και τώρα ο εισηγητής Αρνόλδας Αμπραμαβίτσιους και ο εμπειρογνώμων σας, ο εμπειρογνώμων σας και η γραμματεία της ΕΚΟΝ έρθουν εδώ. Έχουμε τη γνωμοδότηση για κάτι που εν μέρει ήδη συζητήσαμε με τον Αντιπρόεδρο Γιούρκη Κατάινεν. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για μια βιώσιμη Ευρώπη. All right. Ωραία, Αρνόλτα. Πρώτα ε, να σου δώσω το λόγο και ε, μετά θα δώσω το λόγο και σε όσους ε, ζήτησαν το λόγο κατά τη συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να του δώσουμε το λόγο. Τώρα μπορείτε να πάρετε το λόγο. Μπορείτε να το ξαναζητήσετε βέβαια. Αρνόλτα, εσύ πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι. Δεύτερος γύρος της συζήτηση. Και θα ασχοληθούμε με τη γνωμοδότηση αυτή για του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, την οποία είχα την τιμή να εκπονήσω. Ελπίζω να συμβάλλουμε έτσι πολύ πρακτικά ως Επιτροπή Περιφερειών στην εφαρμογή των στόχων αυτών. Πρώτον, ζητήσαμε να εκπονηθεί μια μελέτη. Μας έδωσε πολλά στοιχεία. Επίσης, λάβουμε υπόψη και τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε η Επιτροπή μας και ο ΟΣΑ. όπου διαπιστώσαμε ότι το 60% των ανταποκριτών μας ήδη εφήρμοζαν τους στόχους αυτούς. Ε, βλέπετε εδώ ένα χάρτη της χώρας μου και το Δήμο μου. Αναφέρομαι σε πολλές πρακτικές από το δικό μου Δήμο. Ελπίζω όμως ε, κάτι αντίστοιχο να γίνεται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προπαρασκευή της γνωμοδότησης είχα δυνατότητα να συμμετάσχω στην πλατφόρμα των ε, πολυεμπλεκομένων. Πολύ χρήσιμη ήταν η, η πείρα που αποκόμισα. Είχα οριστεί εκεί εκπρόσωπος της Επιτροπής μας και πολλές προτάσεις αναφέροντας το έγγραφο προβληματισμού. Τώρα λοιπόν περνάμε σε ένα επόμενο βήμα που είναι η γνωμοδότηση. Όπως ξέρετε, η συνάλφος Σύρπα Χέρτελ εργάζεται για μια παρόμοια γνωμοδότηση για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης από πλευράς Επιτροπής ΕΝΒΗ. Ελπίζω οι δύο γνωμοδοτήσεις μας αυτές να βοηθήσουν να εφαρμοστούν οι διαφορετικοί στόχοι εγώ ασχολούμαι με τη διακυβέρνηση των στόχων, την τοπική εφαρμογή τους, ε, την οριζόντια προσέγγιση, ενώ η Επιτροπή ΕΝΒΗ ασχολείται με την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον γενικότερα. Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι δύο νομοδοτήσεις καλύπτουν το θέμα πλήρως και άλλοι υποστηρίζονται. Στην ομιλία μου ήδη, ως εκπρόσωπος του ΕΛΚ, ανέφερα ότι χρειαζόμαστε μία συνολική στρατηγική που να περιέχει τους στόχους, χρονοδιαγράμματα για να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά μέχρι το 2030. Και η πρότασή μας για μία νέα βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη 2030 θα πρέπει να αντικαταστήσει τη στρατηγική μας για το 2020 στα πλαίσια της εφαρμογής και του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαίσιου. Αλλά το νέο στρατηγικό θεματολόγιο για την περίοδο 2019-2024 που αναφέρει τις προτεραιότητες συνδυάζεται με αυτά που ανέφερε και το Συμβούλιο. Αλλά δεν ανέφερε αρκετά για τους, βιώσιμού για τους βιώσιμους στόχους. Αυτό είναι λυπηρό. Καλό τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να έχουν κατά νου τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στο μελλοντικό τους πρόγραμμα εργασιών και στο πρόγραμμα φυσικά της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση εκ των κάτω να συμμετέχουν δηλαδή και τοπικοί και περιφερειακοί φορείς και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη τα οριζόντια όργανα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας για να εντάσσονται οι στόχοι αυτοί σε όλες τις πολιτικές. Για παράδειγμα, στην πολιτική συνοχής. Έτσι, θα διασφαλίσουμε την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη και θα διασφαλίσουμε και την βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις ετήσιες ε, μελέτες ανάπτυξης. Και αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν κατά την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Και το γεγονός ότι κρίναμε την γνωμοδότηση αυτή ομόφωνα στη συνεδρίασή μας, ε, στην εξωτερική συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΚΟΝ στη χώρα μας, στην Λιθουανία, στην, ε, στο Δήμο του Ντρούσκινικε αποδεικνύει ότι όλες οι πολιτικές ομάδες, όλοι οι συνάδελφοι παίρνουν πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και ελπίζω το κείμενό μου να είναι αντικειμενικό και να εκπροσωπεί και να εκφράζει όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιφερειών, όλες τις πολιτικές ομάδες. Ελπίζω ο γνωμοδότηση να βοηθήσει να επιταχυνθεί η ε, παγκόσμια κινητοποίηση για την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης και πάνω απ' όλα ελπίζω να συμβάλλει στην ε, μετατροπή τους από μία απλή διακήρυξη προθέσεων σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας στη γνωμοδότησή μου μέσω τροπολογιών ε, μέσω της συμμετοχής σας στην έρευνα που έγινε και επίσης ευχαριστώ πολύ την ε, εμπειρογνώμονά μου την Τάινα το Βασίλειο από το ΕΛΚΑ και τη γραμματεία της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Σας ευχαριστώ όλους. Ελπίζω η γνωμοδότησή μας να βοηθήσει να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ και συζήτηση. Κύριο Αλόνσο Πλουεγουεσέλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή που εστιάζει στον τοπικό περιφερειακό χαρακτήρα. Ότι πρέπει να ιδιοποιηθούμε εμεί, δηλαδή του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί είμαστε το επίπεδο αυτοδιοίκηση που είναι πιο κοντά ε, και γνωρίζουμε καλύτερα το περιεχόμενο αυτών των στόχων. Όπω ε, υπόθηκε και από άλλε ισπανικέ ε, περιφέρειες αυτή τη στιγμή εκπονούμε στρατηγικά σχέδια για να δούμε πώς μπορούμε στα δικά μας εδάφη, εγώ από τη Μούρθια συγκεκριμένα σας μιλώ, ε, πάνω από 1200 άτομα, 40 οικολογικοί, επιχειρηματικοί, πολιτιστικοί φορεί, φορείς, 400 ε, διοικητικοί υπάλληλοι. Εργαζόμαστε για να δούμε τι θα γίνεται την επόμενη τετραετία με στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, επίκεντρο αυτά που είπαν ο εισηγητής και ο Επίτροπος Πολιτικής Συνοχής. Εάν στη νέα περίοδο προγραμματισμού, τα επόμενα 7 χρόνια, καταφέρουμε τα λειτουργικά επιχειρησιακά αυτά προγράμματα ε, του Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη περιλαμβάνει τη χαμηλή εκπομπές ε, άνθρακα οικονομία, το νερό, την αποχέτευση κτλ. ή ε, την εκπαίδευση και την απασχόληση στο πλαίσιο του ΕΚΤ ή την ανάπτυξη τη υπαίθρου αν τα πετύχουμε όλα αυτά, δεν υπάρχει καλύτερο στόχο ε, ε, για να συνεισφέρουμε και να μην μείνει κανένα πίσω. Ε, συγχαρητήρια για μια κόμφα στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τρενιάντη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική έκθεση, πάρα πολύ σημαντική. Θα ήθελα και εγώ να σταθώ στην ε, πτυχή που έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με την κατάρτιση και αναφέρομαι όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους ε, ενήλικες. Εάν λοιπόν θέλουμε να χτίσουμε μια κοινωνία της επιστήμης, της γνώσης, πρέπει να μεταμορφώσουμε τις κοινωνίες μας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την έρευνα, την ε, μηχανία, την κατάρτιση των γυναικών. Πρέπει να στοχεύσουμε ιδιαίτερα στην μόρφωση των ε, ενηλίκων στη διαβιομάθηση. Ή άλλο κινδυνεύουμε να σκάψουμε ακόμα πιο βαθιά χάσματα στις κοινωνίες μας αν δεν καταφέρουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση που παρουσιάζει τώρα η αγορά της εργασίας. Οπωσδήποτε πρέπει λοιπόν να προβληθεί η εκπαίδευση. Και αν στρέψουμε το βλέμμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που είπαν «Make America Great Again», ναι, οι επιχειρήσεις είναι αυτές που κάνουν θέσεις εργασίας, αλλά και εκατομμύρια είναι αυτοί οι μηχανικοί που κάθε χρόνο αποφυτούν από τα πανεπιστήμια της Κίνας. Άρα πρέπει να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες για απορρόφηση, πρέπει να μιλήσουμε και για τα... Ε, για τις υπηρεσίες της υγείας και ευχαριστώ πολύ. μεγάλη χαρά να λαμβάνω πρώτος ηγητής ε, την ε, εισήγηση αυτή τη γνωμοδότηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, ένα κοινό ε, μια κοινή κληρονομιά θα έλεγα σε σχέση με την επικαιροποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή μας. Βεβαίω ο στόχος της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να χτιστεί η νοοτροπία, ο τρόπος σκέψης που οδηγεί στην αηφορία, στην βιωσιμότητα και δεύτερον πρέπει να μιλήσουμε για την μετάβαση, την ενεργειακή βεβαίω, αλλά και κάθε άλλη μορφή μετάβαση και μεταμόρφωση που έχει το κόστο τη ένα κόστο το οποίο σήμερα μπορεί να ε, χρηματοδοτείται ή να επιδοτείται, να αυτό επί παραδείγματι της ε, ανακαίνησης προς, τον ενεργειακό, προς την ενεργειακή εξοικονόμηση των κτηρίων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μετατραπεί ε, σύν το χρόνο ε, και οικονομικά. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει οι τοπικέ αρχέ, οι περιφερειακές αρχές να ε, αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση οργανώνοντας το νέο σύστημα με την συνεργασία οπωσδήποτε και του ιδιωτικού τομέα των επιχειρήσεων, γενικά του οικονομικού και πιστοτικού συστήματος που θα οδηγήσει στη μετάβαση που θέλουμε εμείς σε τοπικό επίπεδο να υλοποιήσουμε πλέον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω συμπληρώνοντα τη συζήτηση τα συμπεράσματα που αποκομίσαμε από τη χθεσινή συζήτηση. Έγινε μια παρουσίαση, έγινε συζήτηση στη συνέχεια με παρουσία και των πρεσβευτών για το κλίμα από την Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και μετά είδαμε άλλου εκπροσώπους, 20-30 μέλη τη επιτροπή μα, που ήρθαν να συμμετάσχουν μαζί με άλλου, με το ευρύ κοινό θα λέγαμε ε, και άλλους ενδιαφερόμενους ε, με αυτά λοιπόν διαμορφώνονται οι κύριες ιδέες για την προαγωγή του πρεσβευτή περιβάλλοντος της Επιτροπής των Περιφερειών. Είδαμε πολύ καλές ποιοτικέ παρουσιάσεις από την Οβάρα, την ε, Εμίλια Ρωμάνα, τη Γαλλικία και Αρκετές ουσιαστικέ παρεμβάσει ε, από ειδικού, από, ε, από τον Επιτρόπο των ίδιων, από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να αποκόψουμε το κλίμα την κλιματική αλλαγή ως θέμα προς αντιμετώπιση ανήκει στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους διατρέχει. Και εδώ έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία που μας καλεί να προσφέρουμε ιδέες για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του έτους. Κάθε περιφέρεια, κάθε πόλη, με την γύρω Ήπεθρο μπορεί να συμβάλλει στην, στο στόχο αυτό αναπτύσσοντας το δικό της σχέδιο, το δικό της πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας, για την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και επίσης αυτό που τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα είναι ότι πρέπει να γίνει σε επίπεδο πολυεπίπεδου διαλόγου ε, η πρόοδος αυτή, όχι μόνο με την κεντρική κυβέρνηση. Οφείλει η κεντρική κυβέρνηση να παραμένει σε επαφές, σε διαβουλεύσεις να ακούσει τις απόψεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα γίνει βέβαια και η επεξεργασία. Αλλά εδώ μπορώ να πω ότι παρουσίασα τις ε, χθεσινές συζητήσεις και τα όσα είχαν να προτείνουν οι πρεσβευτές κλίματος οι δικοί μας και όχι μόνο για το κλίμα αλλά γενικότερα. Και τώρα αν δεν έχετε αντίρρηση προχωρούμε στην ψηφοφορία με δύο τροπολογίες κάτι μου λέει ότι θα είναι υπέρ ο εισηγητής Υπάριθμον ένα λοιπόν υπέρ παρακαλώ κατά ουδής κρύβεται η δεύτερη τροπολογία υπέρ ευχαριστώ κατά ουδής το σύνολο όπως τροποποιήθηκε υπέρ παρακαλώ κατά ουδής αποχές ουδεμία και εγκρίνεται ομόφωνα κύριε εισηγητά σας ευχαριστούμε πολύ καλή δουλειά σας Thank you. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα. Γνωμοδότηση για την βιώσιμη βιοοικονομία για την Ευρώπη. Ενίσχυση της σύνθεσης οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Ο Γιάσιν Χόρβατ είναι ο εισηγητής μας. Οπότε να του δώσω απευθείας τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι η βιοοικονομία η, δηλαδή η οικονομία που βασίζεται στην βιομάζα σχετίζεται κατά πολύ με τα προηγούμενα θέματα γιατί χωρίς την βιοοικονομία δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης δεν θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ε, υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλάβαμε στο Παρίσι η βιοοικονομία αυτή τη στιγμή έχει κύκλο εργασιών 2,3 δις ευρώ και απασχολεί 8,2 Είναι σημαντικό τμήμα της οικονομίας μας. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να βοηθήσει να εφαρμόσουμε τους στόχους των Παρισίων. Πρόκειται για τον εξυγχρονισμό της ε, βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη και τη δημιουργία νέων αλυσίδων αξία Μία βιώσιμη βιοοικονομία είναι τμήμα της κυκλικής οικονομίας. Τα βιοαπόβλητα μετατρέπονται σε πόρο και οι καταναλωτές θα είναι σε θέση έτσι να μειώσουν κατά 50% τα οικιακά απόβλητα εντός της ε, προσεχούς δεκαετίας. Η βιοοικονομία συμβάλλει επίσης σε ωκεανούς χωρίς πλαστικά. Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης της, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2017. Και αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, παρουσίασε μία ανακοίνωση πάντα για τη βιοοικονομία. Η γνωμοδότησή μας είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτήν την ανακοίνωση της Επιτροπής. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό μέχρι το 2024 κάθε περιφέρεια θα πρέπει να έχει ένα ε, πρόγραμμα, μια στρατηγική. Σε πολλές χώρες αυτό είναι ήδη πραγματικότητα. Πολλές περιφέρειες ήδη έχουν εκπονήσει αυτά τα προγράμματα, αλλά όχι όλες, ορισμένες βραδιπορούν θα πρέπει να λάβουν την επιπλέον ενίσχυση που χρειάζονται και στήριξη για να ε, ανακτήσουν αυτή την καθυστέρηση, να καλύψουν αυτή την καθυστέρηση. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει ένας ενιαίος πίνακα αποτελεσμάτων, ούτω ώστε να έχουμε μετρήσιμού στόχου βιοοικονομίας. Άρα πρέπει να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία και συγκρίσιμοι οι δείκτε, λοιπόν. Για να εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική χρειαζόμαστε ε, υπεύθυνη προσέγγιση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ούτω ώστε όλα τα στοιχεία της στρατηγικής να εφαρμοστούν πλήρως και συνεπώς. η Δήμοι είναι ε, το επίπεδο στο οποίο πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα και πρέπει να έχουμε και συλλογή στοιχείων η βιοοικονομία έλεγα. Χρειάζεται ολιστική προσέγγιση. Γιατί κοιτάξτε, είναι ε, μεγάλης διάστασης μετατροπή αυτό που κάνουμε και η χρηματοδότηση λοιπόν πρέπει να προκύψει από διάφορε πηγέ. Αλλιώ δεν θα είναι επαρκή. Και αν δεν είναι επαρκή. καταλαβαίνετε δεν αρκεί χρηματοδότηση μόνο από το Γεωργικό Ταμείο και το Περιφερειακό Ταμείο. Χρειαζόμαστε και άλλε πηγέ χρηματοδότηση, αλλιώ δεν θα μα φτάσουν τα λεφτά. Πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, βεβαίω, για να υποφευθούν επικαλύψει στην περίπτωση πολλαπλών πηγών χρηματοδότηση. Επίση, πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτη. Να υπάρξει σωστή πληροφόρηση και υπεύθυνη. Το αναφέραμε ήδη σήμερα. Για όλου του τομεί ισχύει, άρα φυσικά ισχύει και την βιοοικονομία. Ενημέρωση λοιπόν του κοινού. Το αναφέρουμε στη γνωμοδότησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας, τις ε, τροπολογίες σας, τη συμβολή σας όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό σε επίπεδο επιτροπής. Με τη βοήθειά σας βελτιώσαμε τη γνωμοδότηση αυτή και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν καθόλου τροπολογίες. Ευχαριστώ την Βαλέρια και την Όλγα για τη βοήθειά τους και επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο Άκοσκόσα τον ε, εμπειρογνώμονά μου. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή γνωμοδότηση και καλύπτει συνολικά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και ο πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Η κυρία Γιώμη Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας για την θαυμάσια εργασία του. Το θέμα αυτό είναι μεγάλη σημασία. Το είπαμε επανειλημμένα σήμερα. Είμαστε φιλόδοξοι. Θέλουμε να επιτύχουμε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050 και τα περισσότερα κράτη-μέλη το στηρίζουν αυτό. Θαυμάσιο αυτό. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο θα πρέπει το Corpus Juris η νομολογία δηλαδή στην Ευρώπη και η νομοθεσία να απλουστευτούν. Γιατί είναι πολύ διαφορετικέ οι αρμοδιότητε για την αντιμετώπιση του θέματο αυτού σε διάφορε χώρε. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, καταφέραμε ουσιώδη πρόοδο. Χρησιμοποιώντα, για παράδειγμα, την, το, την κατανομή τη θέρμανση, τη βιομάζα, τα νέα καύσιμα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάπω επιφυλακτική έναντι όλων αυτών των νέων μεθόδων. Θα έπρεπε να ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για τη βιοοικονομία. Το κριτήριο βιωσιμότητα ε, θα πρέπει να είναι ακριβώ ε, το βασικό κριτήριο για την εφαρμογή τη πολιτική μα. Ε, παρ' όλα αυτά διαπιστώνω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπα, η χρήση τη βιομάζας δημιουργεί κάποιε επιφυλάξει. Τα φορολογικά κίνητρα, για παράδειγμα θα πρέπει να βοηθήσουν, να συμβάλλουν και εκείνα. Ούτω ώστε ε, να προωθήσουμε την καλλιέργεια προϊόντων όπως ε, το έλαιο από κόλζα που μπορεί να βοηθήσει στη βιομάζα. Είμαι λοιπόν επικριτική έναντι τη προσέγγιση της Κομισιόν. Ε, Μα δυσχεραίνει αντί να διευκολύνει την εξέβρεση, την εξέβρεση λύσεων δεν θέλει να εξετάσει τι σωστέ πρακτικέ κάποιων κρατών μελών που όντω έχουν αποδείξει ότι λειτουργούν όπω τα δικά μα. Ελπίζω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζω να είναι κάποιο από εδώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ που να ακούει, ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει, θα απλουστεύσει τη δράση των κρατών μελών για θέματα βιοοικονομία. Γιατί όπω σα είπα, από μικρά ριάκια γίνονται μεγάλοι ποταμοί. Δεν υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Αν όχι, δεν υπάρχουν τροπολογίε. Οπότε να κάνουμε τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Μία. Όχι. Είστε κατά, μάλιστα. Ωραία. Μία ψήφος κατά. Ωραία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Uh, uh, Επόμενη γνωμοδότηση του συναδέλφου Τσάμπα Μπόρμπολ για την ενίσχυση τη διδασκαλία των θετικών επιστημοτεχνολογίας Μηχανική μαθηματικών STEM στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελάτε εδώ παρακαλώ με τον εμπειρογνώμονα και τον εκπρόσωπο τη ε, ΣΕΝΤΕΠ. All uh, uh, Χωρίς ε, άλλη καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον Τσάμπα Μπόρμπολη να μας κάνει την εισαγωγή στην γνωμοδότησή του. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Stimați colegi, stimate domnule președinte, în uh, calitate de raportor al proiectului de aviz... Αξιότιμοι συνάδελφοι, Είμαι εισηγητή τη γνωμοδότηση για την ενίσχυση τη διδασκαλία των θετικών επιστημών, τη τεχνολογία, τη μηχανική των τεχνών και των μαθηματικών, STEAM, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ πω ε, το κείμενο αυτό εδράζεται ε, σε όση συμβολή πήραμε από όλους τους εμπλεκομένους που μας είπαν ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εκπαίδευση ε, ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων. Οι ε, ε, ειδικευμένοι ε, μεταναστεύουν, έχουμε φυγή εγκεφάλων, κάτι που συνιστά μείζον πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πλήττει ιδίω τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στην περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Λύσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός οικονομικού μοντέλου που θα βασίζεται στις γνώσεις και στην ισότητα ευκαιριών. Η Φιλανδική Προεδρία δημοσιοποιεί το πρόγραμμά της σήμερα με επίκεντρο την παιδεία και μετά από πολύ καλή συνεργασία που είχαμε ε, η Ρουμανική και η Φιλανδική Προεδρία νομίζω ότι θα μπορέσει η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και επί Φιλανδικής Προεδρίας ώστε η ευρωπαϊκή εκπαίδευση να είναι καλύτερη στον κόσμο. Αν μου επιτρέπετε τώρα να μιλήσω ουγγρικά από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε ε, τι λύσεις μπορούμε να εφαρμόσουμε και τι λύσεις μπορούμε να βρούμε ώστε να μένουν στη χώρα τους ε, οι άνθρωποι, οι νέοι ιδίω. Το STEM αυτό, η STEAM θέλουμε να το ενισχύσουμε. Θέλουμε να υπάρχει επαφή μεταξύ πραγματικής ζωής και εκπαίδευσης. Θέλουμε τις επιστήμες, ε, τις τεχνικές γνώσεις, τη μηχανολογία, τα μαθηματικά να τα ενισχύσουμε. Πρόκειται για σημαντικούς επιστημονικούς κλάδους ε, ε, και για την οικονομία και για την οικονομική ανάπτυξη. Η δημιουργικότητα έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εξού και πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ε, με τη βοήθεια αυτών, της δασκάς αυτών των αντικειμένων για να μειώσουμε και την ανεργία. Σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις και προβλήματα για να τα υπερπηδήσουν αυτά τα προβλήματα ε, οι, αυτό, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, μπορούν να προωθήσουν ε, τη STEM εκπαίδευση για μεγαλύτερη προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας πρέπει να δώσουμε δουλειά στον κόσμο και ευκαιρίες στους νέους. Αυτό σημαίνει ότι Ορισμένοι φορείς, ορισμένες αρχές και ομάδες ε, διαφερομένων θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και φυσικά και οι τοπικέ και περιφερειακέ περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν ε, γιατί έχουν ένα κρίσιμο ρόλο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε επίσης τη χρηματοδότηση, τι υποδομέ γιατί πρέπει να εστιάσουμε και σε αυτές, όπως και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή των γυναικών. Η δασκαλία των αντικειμένων STEM θα πρέπει να ε, ενισχυθεί και στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης ή τη εκπαίδευση ενηλίκων. Έχουμε στρατηγικέ STEM. Τι εννοώ με αυτό. Ορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να εστιάσουν στις πτυχές που προανέφερα. Επίσης, η δασκαλία STEM θα πρέπει να έχει προτεραιότητα και στο πλαίσιο του προγράμματος Εράσμους και άλλων προγραμμάτων. Επί Φιλανδικής Προεδρίας ε, η κλάδη STEM θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και τώρα να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση, να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Περιφερειών, το ΕΛΚΑ, τη ΣΑΝΤΕΚ, το προσωπικό, Λάς Λότσακ, ένα μεγάλο ευχαριστώ, ε, μεγάλο ευχαριστώ και στην ομάδα ανάλυσης που με βοήθησε. Πρέπει να εστιάσουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτή είναι η άποψή μου. Μόνο έτσι ε, μπορούμε να εστιάσουμε στους νέους παρέχοντάς τους τις κατάλληλες γνώσεις. Και γι' αυτό πρέπει να εστιάσουμε και στους κλάδους STEM. Παρακαλώ λοιπόν να στηρίξετε την γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Παρεμβάσεις υπάρχουν. Καριολάινεν. Πρόεδρε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά αυτή σε ένα θέμα τόσο επίκαιρο. σήμερα και με το πρόγραμμα της Φιλανδικής Προεδρίας υπογραμμίστηκε, υποδημοσιεύθηκε, τονίστηκε ιδιαίτερα το θέμα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του προγράμματος της Προεδρίας της Φιλανδίας. Αν θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε καλή καινοτομία στο μέλλον, εάν θέλουμε ο πολίτης να μπορεί να ωφεληθεί από την καινοτομία, πρέπει να ενισχύσουμε τις δεξιότητες στα τομείς αυτούς ε, των STEM και βεβαίως χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες σε τεχνικά επαγγέλματα άρα χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση και των κοριτσιών στα STEMs αυτά. και έτσι μπορούμε να έχουμε πρέπει να δώσουμε καλύτερα έμφαση ήδη από το δημοτικό από την τρίτη τετάρτη δημοτικού όταν αρχίζει το παιδί να ενδιαφέρεται για τα φυσικά φαινόμενα στα μαθήματα αυτά των θετικών επιστήμονων που βέβαια χρειάζεται να έχουμε και εμπνευσμένου καθηγητές αλλά και σχολεία με άριστες υποδομές. Αυτά μπορούν να τα εξασφαλίσουν οι τοπικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη δουλειά. Μετά τη Ρουμανία αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση στο Συμβούλιο και στο σκοπεύουμε και εμείς να παραγάγουμε την διδασκαλία των STEMS. Ευχαριστώ πολύ Κόμπορ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση από την γνωμοδότηση που μελέτησα. Ε, είμαι καθηγητής φυσικός και διαπιστώνω στον επαγγελματικό μου βίο πως υπάρχουν τεράστια κενά μεταξύ των αναγκών και της γνώσης της επιστημονικής. Και διαπιστώνω επίση ότι όποιο δεν έχει επαρκή επιστημονικέ γνώσει δεν μπορεί να βρει μια θέση στην αγορά εργασία ε, καλή, δεν μπορεί να διαχωρίσει, φερειπίνη για την κλιματική αλλαγή, τι είναι επιστημονική ε, έκθεση και πρόβλεψη και τι είναι λαϊκιστική ε, θέση και είδηση ψευδής και βεβαίω πρέπει να ενισχυθούν τα STEM σε όλα τα σχολεία. Τα σχολεία όμω είναι διαφορετικά στην Ευρώπη. Παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με την διδασκαλία των θετικών επιστημών. Σε ορισμένε χώρε, όπω στην Ουγγαρία, παραδείγματι, έχουν ε, ε, τα δευτεροβάθμια, τα γυμνάσια και τα λίγα δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάγεται στην κεντρική κυβέρνηση και άρα δεν μπορεί να παρέμβει η τοπική και περιφερειακή κυβέρνηση και επίσης εσωτερική αντίφαση άλλη αυτή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε έχει λόγο στον οδηγό σπουδών η εκκλησία ίδια. Μάλιστα λέει ο πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Αρέστρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συνάδελφος πριν από λίγο μίλησε για την ε, ε, σπάνιδα των κοριτσιών στις θετικές επιστήμες. Βεβαίως, Είναι πραγματικό το πρόβλημα ότι ορισμένε εκπαίδευτε δεν ενδιαφέρονται για τι θετικέ επιστήμε και νομίζω ότι πρέπει αρκετά νωρί να τι πλησιάσουμε για να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον του. Και το ίδιο και χειρότερο πρέπει να πω είναι το φαινόμενο στην ψηφιοποίηση. Έχουμε πολλά λοιπόν να κάνουμε, οφείλουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε. Η ψηφιοποίηση, η καινοτομία απαιτούν και να δούμε τα πράγματα με μια προοπτική φύλου. Πρέπει, πλέον και οι γυναίκες να μπορέσουν να αντλήσουν τα ωφέλη της ψηφιοποίησης. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ε, επιστήμες πρέπει να προχωρήσει με ένα πρόγραμμα δράσης ανοιχτό προς όλα τα παιδιά που θα καλεί, θα προσκαλεί όλα τα παιδιά και θέλουμε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο και στα κορίτσια και γενικότερα στο σχολικό βίο για να μπορεί ο καθένα να συμμετέχει στις εξελίξεις τεχνολογίας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα προχωρούμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία μία. Την ψηφίζουμε. Ο εισηγητή είναι κατά τροπολογία πρώτη λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ κατά. Καταψηφίστηκε το σύνολο της εκθέσεως παρακαλώ όπως έχει υπέρ κατά ουδείς εποχές δεν υπάρχουν και ομόφωνα εγκρίνεται η έκθεση συγχαρητήρια στον κύριο Βόρμπουλη Ωραία. Τώρα θα συζητήσουμε τη γνωμοδότηση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ο συγκριτής μας είναι ο Ούνο Ζίλμπεργκ με τον εμπειρογνώμονα και εκπρόσωπο της Επιτροπής ΝΑΤ. Παρακαλώ. Ωραία. Και τώρα ε, ο κύριος Συγητής. Ευχαριστώ πολύ. Έχω την τιμή να ε, παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειών το θέμα βέβαια μας έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά έχουμε προσθέσει τώρα μία νέα διάσταση. Παρακαλώ, μπορεί να μας πει κανείς αν ήξερε ε, πριν από σήμερα ή πριν από τον τελευταίο καιρό την επιβλαβή επίδραση των ενδοκρινικών διαταρακτών. Αλλά επειδή το συζητήσαμε στην ΑΤ, πολύ μάθαμε. Θεωρώ όμως ότι καλό είναι να σας παρουσιάσω μερικά σημαντικά γεγονότα γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και γιατί πρέπει να ασχοληθούν και οι τοπικές αρχές με την αντιμετώπιση τους. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικό ότι παρουσίασε αυτή την πρωτοβουλία και δεν θα πρέπει να πράξει καμία περαιτέρω καθυστέρηση για την εκπόνηση μιας νέας στρατηγικής για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Επίσης, αυτή η νέα στρατηγική θα πρέπει να συμπληρωθεί με ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με βάση νέα κριτήρια για το τι είναι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες που θα πρέπει να περιέχονται σε όλα τα νομοθετήματα της Ένωσης όπου θα πρέπει για να μεθεί η έκθεση σε τέτοιους διαταράκτες ιδιαίτερα ε, η έκθεση των πιο ευαλώτων τμήματων του πληθυσμού. Το πρόβλημα είναι ότι η ευαισθητοποίηση για το ρόλο που μπορούν να παίξουν αυτοί οι διαταράκτες του κοινού είναι πολύ περιορισμένη. Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν ούτε καν τις έννοιες τι είναι η λειτουργία των ενδοκρινών αδένων και πώς μπορεί να διαταραχθεί. Άρα είναι σημαντικό να υπάρξει περισσότερη ευαισθητοποίηση. Επίσης ε, να αντιμετωπιστεί και η διαφοροποίηση των κανόνων από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των ορισμών και της νομοθεσίας για τις ουσίες αυτές. Αλλά κυρίως πρέπει να φροντίσουμε την υγεία των συμπολιτών μας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και του καταναλωτή και της οικονομίας. Αλλά αν υπάρχει αντίθεση μεταξύ των συμφερόντων της οικονομίας ή κάποιων ε, κλάδων της και από τη μία και των συμπολιτών μας από την άλλη φυσικά η δημόσια υγεία είναι το πρώτο μέλημά μας και δεν είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη σχέση των διαταρακτών αυτών με κάποιες διαταραχές ακριβώς αλλά και με το ρόλο που παίζουν για τα προβλήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον και στα άγρια ζώα γενικότερα δηλαδή στην κοινωνία πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι πρέπει να είναι και σαφές το μήνυμά μας. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να είναι διατεθειμένες να προστατεύσουν τις μελλοντικέ γενναίες. Παρά την πίεση, για παράδειγμα, από ισχυρές ομάδες ε, πιέσεων και από κάποιους εμπορικούς μας εταίρους. Το θέμα αυτό, όπως σας είπα, βεβαίως είναι και πολύ παλιό, αλλά παράλληλα και πολύ επίκαιρο. Και στο σχέδιο γνωμοδότησής μου, όλα αυτά τα θέματα με όλα τα υποθέματα έχουν παρουσιαστεί λεπτομεριακά. Οπότε, ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στη συζήτηση, υπέβαλαν τροπολογία στην Επιτροπή ΝΑΤ και επίσης ευχαριστώ τους συναδέλφους μου γενικά από την Επιτροπή αυτή και να ευχαριστήσω και τον καθηγητή Άντερς Βάλτμαν που ήταν ο εμπειρογνώμονας μου και συνέβαλε πολύ στην εκπόνηση του κειμένου μου που είναι τόσο αναλυτικό, αλλά παράλληλα ισορροπημένο και αντικειμενικό. Μόνο μία τροπολογία έχει υποβληθεί και νομίζω ότι θα περάσουμε στη συζήτηση για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν μία τροπολογία, αλλά θέλει κανείς να πάρει γενικά το λόγο από αυτού του θέματος. Όχι. Οπότε περνάμε στην ψηφοφορία επί της τροπολογίας. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Κανείς. Ωραία, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποιηθή σε γνωμοδότηση υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές ούτε κατά ούτε αποχή ομόφωνα εγκρίνεται. Συγχαίρουμε τον εισηγητή μας. Right, so... Καλώς. Αυτές ήταν οι γνωμοδοτήσεις μας για σήμερα. Και αύριο έχουμε μερικές προς ψήφιση. Αλλά σήμερα το επόμενο θέμα είναι τα ευρωπαϊκά θέματα της τοπικής αρχές. Όπως ξέρετε, στις δύο προηγούμενες ολομέλειες συζητήσαμε παρόμοια θέματα όπου εκ των προτέρων ζητάμε από τα μέλη μας αν θέλουν να υποβάλουν προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση. Με βάση μία σύντομη αιτιολόγηση και κατόπιν η διάσκεψη των Προέδρων επιλέγει τα θέματα που θα συζητηθούν. Είχαμε επιλέξει λοιπόν δύο θέματα αρχικά, αλλά δυστυχώς ε, λόγω της απουσίας των συναδέλφων που τα πρότειναν θα συζητήσουμε μόνο ένα είναι η διαδικασία κοινοποίησης για τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Οπότε να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Πέτα Κούατς για να μας πει πώς η κατάσταση αυτή επηρεάζει την πόλη σας. Και, και μετά θα μας ενημερώσει και ο κύριος Γιόγκμαν από την Ολλανδική Αντιπροσωπεία που θα μας παρουσιάσει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες. Άρα ίσως ε, δεν είναι παρόν, ίσως κάποιος άλλος από την Ολλανδική Αντιπροσωπεία θα τον αντικαταστήσει. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τον Πέιτα Κούρτς. Και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο και στους συναδέλφους τον το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που θέσατε το θέμα στη μέση διάταξη. Θα ήθελα να το διευκρινίσω λίγο. Αφορά όχι μόνο τις κατοχώρες και τη Γερμανία, τις δικές μας χώρες, αλλά πολλές κοινότητες και δήμους στην ε, Ευρώπη. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με την οδηγία για την κοινοποίηση, αλλά γιατί, για το ότι χάρη στην οδηγία αυτή μπορούμε να ξεπεράσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ουσιαστικό. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με, ένα, με μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2018, του Ιανουαρίου του 2018, μέχρι την οποία θεωρούνταν γενικά από όλους ότι τα ρημοτομικά σχέδια δεν υπάγονται, αυτά δηλαδή που εκδίδουν οι Δήμοι, δεν υπάγονται στην οδηγία για την παροχή υπηρεσιών. Αποφασίζει όμως το δικαστήριο ότι ενδέχεται να υπαχθούν εφόσον μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της δραστηριότητας του ε, εμπορίου. Άρα, όταν έχουμε ένα ρηματομικό σχέδιο σε μία πόλη και ενδεχομένως προσφορά εμπορικών ε, δραστηριοτήτων που μπορεί να σχετίζονται με το κέντρο μιας πόλης ε, ε, μπορεί να αποκλειστούν από την λειτουργία τους στο κέντρο αυτό της πόλης, φερειπίν βιοτεχνικές δραστηριότητες ή βιοτεχνικές περιοχές και όλα αυτά ενδέχεται τότε να υπάγεται στην ε, οδηγία περί παροχής υπηρεσιών και άρα κάθε τέτοιου ε, είδου σχέδιο, κάθε ρηματομικό θα πρέπει πλέον να υποβάλλεται και να κοινοποιείται για ε, επιβεβαίωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ μιλούμε για χιλιάδες δήμους με εκατοντάδες ρηματομικά ή αντίστοιχα σχέδια το χρόνο. Αυτό σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες διαδικασίες κοινοποίησης μόνο από τη Γερμανία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με τεράστιο γραφειοκρατικό όγκο αλλά και με άρνηση της ε, βασικής αρχής σε πρωτογενές επίπεδο ε, παραγωγής νομοθετικής ε, πράξης από τους Δήμους, τα αρωματομικά του σχέδια δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε να περιοριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να το αποδείξει ότι ασχολείται μόνο με τα θέματα τα οποία πραγματικά μπορεί καλύτερα να λύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην παρεμβαίνει κατά τρόπο παρεμποδιστικό ή και καταστροφικό ακόμη μερικές φορές σε τόσο ε, τοπικό επίπεδο. Κάτι το οποίο προκύπτει σαν αποτέλεσμα και ότι κανείς δεν είχε την πρόθεση να υπαγάγει τα ρημοτομικά αυτά σχέδια ή τα σχέδια των ε, Δήμων στην οδηγία περί παροχής υπηρεσιών. Εννοείται ότι δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί μέσω του Κοινοβουλίου η ε, νομολογία του δικαστηρίου και μόνο εάν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια νέα πρωτοβουλία, πρωτοβουλία από το Κοινοβούλιο μεν αλλά και από το Συμβούλιο για μια νέα νομοθετική παρέμβαση, γιατί μόνο αυτό θα μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση, μια κατάσταση η οποία θεωρώ πως μπορεί να έχει τεράστια ε, συνέπειες και θα αποβεί εις βάρος γενικά των τοπικών και δημοτικών αρχών, αλλά και γενικότερα της Ευρώπης. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ κύριος Δεχέρ, η ε, Ολλανδική αντιπροσωπεία παρακαλώ, κατοχώρηση. χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη γραμμή του Γερμανού συναδέλφου και θα τον υποστηρίξω. Παρακολουθούμε την Κομισιόν από όταν έκανε την πρώτη παρουσίαση το 2017 ο άδελφο Φαντεράς είχε κάνει μια πάρα πολύ ωραία νομοδότηση. Η οδηγία λοιπόν για την κοινοποίηση ε, διευρύνει την υποχρέωση κοινοποίηση. Υπάρχει περίοδος διαβούλευσης τριών μηνών. Και υπάρχει που σημαίνει δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Δηλαδή τα σχέδια που αποφάσισαν τοπικές ή περιφερειακές αρχές και έχουν ήδη μελετηθεί μπαίνουν στο ψυγείο κατά κάποιο τρόπο για τρεις μήνες. Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή τους. Και για να μην παρεξηγήσει κανείς, δεν είμαι κατά της παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν θέλουμε διοικητική επιβάρυνση, διοικητικό άγχος, άχθος, αλλά πιο μεγάλη σαφήνεια ε, σε αυτά τα χωροτοξικά σχέδια. Με αυτή την ασάφεια ε, δυσκολεύει, ε, δυσχεραίνεται η ζωή και των τοπικών αρχών και των πολιτών εν γέννη. Πρέπει τώρα όμως να βρούμε όλοι μαζί μια λύση και γι' αυτό παρακαλώ όλα τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών όπως και ο κύριος Κούρτς, απευθύνω και εγώ έκκληση να μιλήσουμε και στους αρμοδίους σε εθνικό επίπεδο για να λυθεί το πρόβλημα και πρέπει να μείνει προτεραιότητα το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει άλλο στο λόγο. Αν όχι, ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος αυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το θίξατε το θέμα αυτό. Επόμενο θέμα. Στην ημερήσια διάταξη. Η Ευρωπαϊκή, τα βραβεία για την ευρωπαϊκό ε, επιχειρηματικότητα. Και καλωσορίζουμε λοιπόν την ε, σχετική επιτροπή και τους ε, που έχουν ε, ήδη ενημερωθεί. Τρεις είναι οι νικητές. Έχουμε και κάποια μέλη ε, της Επιτροπής ε, Επιλογής. Αν θέλετε λοιπόν να έρθετε για να κάνουμε τις συζητήσεις. Το πρόγραμμα αυτό για τις ε, περιφέρειες ε, επιχειρηματικότητας πλέον έχει κλείσει 10 χρόνια ύπαρξης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να απονείμω τα βραβεία αυτά μιας και συμμετείχα από την αρχή. Με τη δική μου την περιφέρεια στο Ελσένκι, Ότσιμα και βραβεύτηκε η περιοχή αυτή. Και πρόσφατα ήμουνα ε, πρόεδρος της ε, Επιτροπής να σας πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η επιλογή των περιφερειών. Ιδιαιτέρως ε, φέτος με τον κατάλογο των περιφερειών που είχαν υποβάλει υποψηφιότητα με λεπτομερείς ε, προτάσεις. Αυτό πραγματικά καταδεικνύει πόσο υψηλή ποιότητας είναι οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Και επίσης ε, όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ήθελαν να δουν και τι κρύβεται πίσω από το κείμενο της υποψηφιότητας. Εξέτασαν λοιπόν όλες τις περιφέρειες αντελεχώς και είμαστε απόλυτα πεπισμένοι λοιπόν στην τελική απόφαση που λάβαμε σε ό,τι αφορά τους τρεις νικητές. Πρωτού επισέλθω σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρεια, να καλέσω του εκπροσώπου των περιφερειών να ανέβουν εδώ. Γκτάνσκ, Πομόρσκι. Uh, Έχουμε και το Gothenburg της Σουηδίας η επιχειρηματική περιφέρεια και στη συνέχεια έχουμε και την ε, Λαμάρα από την Ισπανία. Uh, Παρακαλώ, περάστε. So we have here, uh, uh, first, uh, from, Να ακούσουμε πρώτα την ε, περιφέρεια Πομόρσκι. Ο Μίτσισλαβ Στρουκ. Τον γνωρίζουμε πολύ καλά. Καλώς ορίσατε με τον αντιδήμαρχο της, ε, του Ντάνσκ, τον κύριο Αλεξάνδροβιτς. Καλώς ορίσατε. Άξελ Γιούζεφσον, πρόεδρο, ε, μάλλον πρόεδρος της, ε, των τοπικών περιφερειών του Γκέτεμπορκ και επίσης πρόεδρο της εκτελεστικού συνεδρίου της Πόλεως, του Δήμου. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Μάνο Αγιάρντη, αντιπρόεδρο της ε, κυβέρνησης της Ναβάρα. Να σας πω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη κακαλιά και την κινητήριο μηχανή της οικονομίας και σε αυτή τη δέκατη επέτειο των βραβείων βλέπουμε μια τεράστια πρόοδο σε ό,τι αφορά τις ε, νεοφυεί επιχειρήσεις, το πώς διαμορφώνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς έχουν διδαχθεί ουσιαστικά οι περιφέρειες η μία από την άλλη. Αυτό αποτελεί ένα καλό τεκμήριο για την ιδιαίτερη σημασία που φέρει αυτό το βραβείο. Γιατί έχουμε διάφορες τάσεις, παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση, αλλαγές στην συμπεριφορά των καταναλωτών. Όλα αυτά τα επόμενα χρόνια θα αναγκάσουν τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ορίσουν εκ νέου τις δραστηριότητες του, σε ό,τι αφορά και τις τοπικές δραστηριότητες τους. Για παράδειγμα, ε, τοπικές βιομηχανίες, πανεπιστήμια, όλοι αυτοί θα πρέπει να προσαρμοστούν και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης θα καθοριστεί από τον τρόπο που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας θα ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Προκειμένου να πετύχουν θα χρειαστούν ένα επιχειρηματικό προφίλ με ανάλογες ικανότητες και ανάλογη εμπειρία προκειμένου να διαμορφώσουν και αυτές ε, την κοινωνία και την οικονομία. Έχουμε θέσει λοιπόν μια πενταετή περίοδο προτεραιοτήτων. Έχουμε ζητήσει βιώσιμη ανάπτυξη και ζητούμε επίσης διαδικασίες bottom από, πάνω, από κάτω προς τα πάνω. Τονίζουμε τα τρία κριτήρια που θέλουμε να υπάρχουν, να υπάρχει σωστή πρόοδος και ο Καλ Χάινς Λάμπερτς και εγώ Έχουμε εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Το πρώτο από τα τρία αυτά κριτήρια είναι ε, μια νοτροπία επιχειρηματικότητα. Ψηφιοποίηση και έξυπνη εξειδικεύση, τα άλλα δύο κριτήρια. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα τα οποία εξετάσαμε από πλευρά ε, τη Επιτροπή μα. Και καταδεικνύεται λοιπόν ότι οι περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργώντας τις συνθήκες για να υπάρχει ένα πραγματικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας στο οποίο οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς θα συνεργαστούν με παραγωγικό τρόπο, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα. Αυτή η Silicon Valley σε τοπικό επίπεδο λοιπόν, ας την πούμε έτσι, όχι φυσικά αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μας ε, δίνει ευρωπαϊκά μαθήματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Θα πρέπει λοιπόν να, να περάσουν όλα αυτά σε ένα νέο επίπεδο. Η επιχειρηματικότητα λοιπόν σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να περάσει σε άλλο επίπεδο και θα πρέπει να υπάρξει και ανανέωση φέτο του συστήματο ε, μπράβευση τη επιχειρηματικότητα. Αυτό λοιπόν θα ανακοινωθεί επίσημα γιατί η Επιτροπή συνεργαζάνεται και με τη Γενική Διεύθυνση ανάπτυξη, η DG Grow και διοργανώνει και ειδικό συνέδριο σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσεις ε, τέλη Νοεμβρίου στο Ελσίνκι 25 με 27 Νοεμβρίου σε συνδυασμό με την ε, με συνεργασία με την πόλη του Έσπορν. Και εκεί θα ανακοινωθεί λοιπόν επίσημα α, είναι αυτή μορφή και θα ζητηθούν προτάσεις. Κάποιες από τις προτάσεις είναι πολύ καινούριε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που στους νικητές συγκαταλέγεται και η Σουηδία Άρα ο χάρτης της Ευρώπης πλέον είναι πιο ισορροπημένος. Κοιτάμε και κάποιες άλλες χώρες, περιφέρειες που θα καταθέσουν προτάσεις και υποψηφιότητε τις επόμενες φορές και είμαι πεπισμένος ότι αν και κάποιες περιφέρειες δεν ε, επιλέχθηκαν στις τελευταίες ε, βραβεύσεις. Ε, θα είμαστε πολύ ευτυχείς εάν ξανεποβάλλουν τις προτάσεις τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα στο σημείο αυτό να απονείμω τα βραβεία. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο και τον κύριο Αλεξάνδροβιτς για την περιοχή Γκτάντς Κντάνς-Πομορφκή. You're here, uh, Polish. Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω τα πολωνικά. Το βραβείο Περιφερειακής Επιχειρηματικότητας για το 2020 είναι μια μοναδική διάκριση Θεωρούμε ότι αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών μας. Yes, for the TV and other media. Okay, you can continue. Thank you, thank you, thank you. Some words I repeat Nagroda έλεγα λοιπόν, το βραβείο Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ευρωπαϊκής είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το ξεχωριστό. Θεωρούμε ότι αποτελεί επιστέγμα των προσπαθειών μας ενό οράματο που η τοπική και περιφερειακή μας ε, αυτοδιοίκηση προσπάθησε να επιτύχει με την περιφερειακή τη στρατηγική ανάπτυξη. Είμαστε υπερήφανοι που ηγούμαστε ως περιφέρεια όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τομείς της οικονομίας. Έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχουμε καταφέρει να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις στην περιοχή μας και είναι εξωστρεφής η οικονομία της περιοχής μας. είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να προσαρμόζεται στις αλλαγές, να επιδεικνύει ευελιξία. Είναι μία από τις προκλήσεις των καιρών μας. Το γεγονό ότι υπάρχει όλο και πιο μεγάλος ανταγωνισμός για την προσέλκυνση ταλαντούχων ε, ανθρώπων. Στο Γκτάνσκ προσπαθούμε να προωθήσουμε τη διαφορετικότητα και ο συνάδελφος που εκπροσωπεί την περιφέρειά μας και ο οποίος Αντάμοβιτς ε, έχει ε, παρευρεθεί σε κάθε συνάντηση και σε κάθε ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών. Θεωρούμε ότι το βραβείο αυτό αντικατοπτρίζει τα δυνατά στοιχεία, δυνατά σημεία της περιφέρειάς μας, και την προσήλωσή της στις ευρωπαϊκές αξίες. Θα θυμάστε ιστορικά πώς δημιουργήθηκε ο οικισμός στην περιοχή του Γκτάνσκ. Έχουμε ε, πρόκειται για μια κοινότητα η οποία βασίστηκε στο εμπόριο. Και αυτή η φιλοσοφία ε, τη συνεχίζουμε. Το ξεχωριστό αυτό βραβείο λοιπόν Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικότητας είναι ένας τρόπος και εμεί να επαναβεβαιώσουμε την δέσμευσή μας, να προσπαθήσουμε όχι μόνο για την, να προωθήσουμε την ε, οικονομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά επίσης και να δημιουργήσουμε δίκαιες συνθήκες ε, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της περιοχής μας να υποφελούνται από την ανάπτυξη αυτή, συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η δεύτερη απονομή. Α, όχι, θέλει και ο κύριος Αλεξάνδρος το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τιμή για μένα που παρευρίσκομαι και θα ομιλήσω στην Πολωνική. Είμαι πολύ υπερήφανος που η πόλη του Γκτάνσκ και η περιφέρεια του Πομόρσκι βραβεύτηκε για το επιχειρηματικό πνεύμα το οποίο επέδειξε για το 2020. Αυτό αποδεικνύει ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν τα έχουμε χάσει στην Πολωνία και επίσης τα 15 χρόνια που είμαστε μέλη της Ένωσης τα εκμεταλλευτήκαμε σωστά. Το Γκτάνσκ είναι η πρωτεύουσα της περιοχής Πομόρσκη είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα, επηρεάζει το σύνολο της περιφέρειας σε πολλούς τομείς μεταξύ των οποίων και την επιχειρηματικότητα. Εδώ και αρκετά χρόνια ε, είχαμε θέσει ένα πολύ σημαντικό στόχο να προσελκύσουμε στην περιοχή μας τους πιο εκλεκτούς επιχειρηματίες οι οποίοι σέβονται το περιβάλλον, σέβονται την κληρονομιά μας, ε, επιδεικνύουν ε, δημιουργικότητα, φαντασία ανεξαρτήτως της ηλικίας του φίλου ή της θρησκείας, του σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή ό,τι άλλο. Αν δει κανείς τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, έχω την αίσθηση ότι τους περισσότερους στόχους μας τους πετύχαμε. Το Gdansk σήμερα δεν είναι μόνο ένα μέρος το οποίο αναπτύσσεται η παραδοσιακή οικονομία και αναφέρομαι στην ναυτική βιομηχανία ή στα καύσιμα αυτό το οποίο μας καθιστά ε, ξεχωριστούς ε, είναι το πρωτοποριακό μας πνεύμα. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε ε, όλους τους ανθρώπινους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και να επανέλθουμε στην παράδοση του χανσεατικού συνδέσμου Συνειδητοποιώ λοιπόν την δυνατότητα αυτή που έχει η περιοχή να επηρεάσει τις οικονομικές εξελίξεις. Αυτά όλα καθιστούν το Γκτάνσκ ξεχωριστό. Αυτό επίσης καθιστά το Γκτάνσκ ξεχωριστό και σε τομέα διοίκησης, επιχείρησης, κοινωνικής οργάνωσης κτλ. Το όραμά μας αυτό γίνεται πραγματικότητα δημιουργούνται νέα μοντέλα ενσωμάτωσης των μεταναστών Θέλουμε να βοηθήσουμε το Γκτάνσκ να αναπτυχθεί σωστά, να είναι ένα σωστό μέρος για να ζει κανείς, ένα μέρος που εμπνέει, που δίνει ενέργεια, δίνει πάθος, ε, αλλά ταυτόχρονα είναι σύγχρονο και δεν ξεχνά το ιδιαίτερο παρελθόν του. Επιμένουμε στα πολιτιστικά θέματα, επενδύουμε στην παιδεία, στον αθλητισμό, στο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην σωστή ποιότητα της ζωής των πολιτών μας. Υπάρχει μια καλή αγορά στον τομέα της κατοικίας, ο τουρισμός είναι σημαντικός, αν δει κανείς ότι το 18 δεχθήκαμε 3 εκατομμύρια επισκέπτες και απασχολούνται πάνω από 3.000 ε, εργαζόμενοι εκεί. Συνεπώς λοιπόν το Γκτάνσκ είναι εκεί, είναι παρόν, είναι εύκολο να πάει κανείς, ε, συνδέεται με τις υπόλοιπες πόλεις της Πολωνίας είτε αεροπορικά είτε με ε, οδικό τρόπο ή και με πλοία. Όταν πάει κανείς στο Γκτάνσκ βλέπει ότι αξίζει τον κόπο να μείνει και να το δει και να δώσει ακόμα περισσότερο χρόνο για το μέλλον της περιοχής. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι το βραβείο αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμα κίνητρο και θα μας καταστήσει ικανούς να εκμεταλλευτούμε καλύτερα το επιχειρηματικό μας πνεύμα για την πόλη μας, την περιφέρειά μας και τη χώρα μας. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους που είναι παρόντες. Χάρη στην προσπάθειά τους πήραμε το βραβείο. Okay, and let me just very briefly... Πολύ σύντομα λοιπόν και εγώ να εκθέσω περιληπτικά το σκεπτικό της Κριτικής Επιτροπής με βάση το οποίο εδώ το βραβείο στο Πιτάνς Μόρσκι γιατί ανέλαβε λοιπόν αυτή η περιφέρεια στοχευμένες δράσεις για την προσέλκυση ικανού προσωπικού, την δημιουργία νεοφιών επιχειρήσεων και φρόντισε για την παροχή ε, υψηλή ποιότητα εκπαίδευση τους νέους. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε, αυτό θέλουν να μάθουν και οι άλλες περιφέρειες πώς να το πράττουν και ελπίζω να έχουμε όλο και μεγαλύτερη συνεργασία, όλο και πιο ισχυρή συνεργασία μαζί σας. Ας περάσουμε τώρα στην περιφέρεια του Κέτεμπεργκ. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Ιώσεφσον, να τονίσω και εδώ τα βασικά στοιχεία που θεωρήσαμε ε, ελκυστικά στην ε, αίτησή σας. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονό ότι έχετε αναπτύξει μια πακροπρόθεσμη στρατηγική σε πολλά επίπεδα, έτσι ώστε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα, να δημιουργηθούν καλύτερε συνθήκε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και θα απονείμε το βραβείο στον κύριο Ιώσεφσον. is yours. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και είμαι ιδιαίτερα περήφανο και ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ σήμερα το απόγευμα και που λαμβάνω το βραβείο αυτό το Γκότεμπορκ. Πολλοί από εσά να μην γνωρίζετε την πόλη του Γκότεμπερκ αλλά δημιουργήθηκε το 1621 και έχει μακρά ιστορία εμπορίου. Σήμερα ωστόσο περιλαμβάνουμε πάνω από 750 βιομηχανίες, ε, κλάδους ε, στην ε, περιοχή του Γκότεμπορκ, από εμπορία μέχρι δομές πολλοτομιακές. Έχουμε πολλά λοιπόν θέματα. Είμαστε στη Βυτική Σκανδιναβία, όπω την αποκαλούμε. 70% της συνολική βιομηχανία βρίσκεται σε 500 χιλιόμετρα απόσταση από το Γκέτεμπορκ. Μιλάμε λοιπόν για μεγάλο κέντρο, για πολλές βιομηχανίες. Έχουμε το μεγαλύτερο λιμάνι στη Σκανδιναβία, μεταξύ Ατλαντικού και Βαλτικής. Περίπου 500.000 σκάφη έρχονται στο λιμάνι μας κάθε χρόνο. Πάνω από 30% των ε, εξαγωγών και εισαγωγών της Σουηδίας περνούν από το λιμένα του Γκέτεμπορκ. Μιλάμε για μεγάλο λιμάνι λοιπόν, το οποίο είναι και πολύ σημαντικό για μας. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε και την ε, σύνδεση με το Όσλο και την Νορβηγία και με την Κοπεχάγη και το Αμβούργο προκειμένου να είμαστε πιο καλά εξοπλισμένοι για τις ανάγκες των επιχειρήσεών μας. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Gothenburg είναι ότι έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Volvo και Είμαστε μοναδικοί στην περιοχή του Gothenburg και οι μοναδικές αρμοδιότητες που έχουμε στην περιοχή σε ό,τι αφορά τη μετάβαση των βασικών βιομηχανιών όπου περνάμε από τα προϊόντα μηχανικής σε προϊόντα κομπιούτερ ουσιαστικά υπολογιστών. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή για μας. Παρά το γεγονό ότι είναι καλά το επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή του Γκότεμπεργκ, διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται και μια στρατηγική για το επιχειρηματικό κλίμα, για την επιχειρηματικότητα, όπω είπε ο κύριο Πρόεδρο και η επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό σημείο για να υπάρξει επιτυχία στο μέλλον και είναι σημαντικό λοιπόν να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή και γι' αυτό λοιπόν αναπτύσσουμε νέες στρατηγικές για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και για να υπάρχει μεγαλύτερο κλίμα επιχειρηματικότητας. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο στόχος να υπάρξουν πιο πολλές από 120.000 νέες θέσεις απασχόλησης μέχρι το 2035 στην ευρύτερη περιοχή του Γκότεμπορκ. Το μοναδικό λοιπόν σημείο που το μοναδικό, αν θέλετε, το ιδιαίτερο πλεονέκτημα είναι η δομή από κάτω προς τα πάνω που ακολουθούμε. Έχουμε πάνω από 40 εργαστήρια, πάνω από 100 επιχειρήσεις ε, συμμετείχαν σε αυτές τις εξελίξεις και αυτό μας οδήγησε σε βασικές ε, σε βασικά επιτεύγματα για να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό κλίμα και να βελτιώσουμε και τις συνθήκε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί φυσικά στοιχείο δηλαδή Μια κρίσιμη πτυχή σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της στρατηγική στην επιχειρηματική κοινότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την επιχειρηματική περιοχή και επιτροπή του Γκέτεμπορ και τη σκληρή δουλειά που έκανα για να πετύχει αυτό. Ιδάλλω δεν θα είχαμε καταφέρει τέτοια αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτό το βραβείο αποτελεί μια επιβράβευση τη δουλειά που κάναμε όλοι μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε για να πετύχουμε ένα σωστό επιχειρηματικό κλίμα, ένα ευνοϊκό κλίμα. Έχουμε μία από τι καλύτερε στρατηγικέ για την επιχειρηματικότητα, θεωρούμε. Αυτό το βραβείο είναι σημαντικό για μα. Θεωρούμε ότι αποτελεί μία απόδειξη για το ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Σα ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ, Άξελ Περνάμε στην περιοχή της Ναβάρας. Σύντομα θα αναφερθώ στα βασικά σημεία της υποψηφιότητάς σας υποδειγματική στρατηγική για τον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών στοχευμένες δράσεις που ενισχύουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις το περιφερειακό σχέδιο επιχειρηματικότητας όπως και η ευφυής εξειδίκευση ήταν και είναι για σας οι βασικοί τρόποι εφαρμογής των στόχων αυτών για τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε όλοι να μάθουμε από τις δικές σας εμπειρίες και γι' αυτό θα σας δώσω κυρία Γιάρδη το βραβείο. Arratsaldeon, Arratsaldeon eskualdetako lantalde lehendakari jauna. Λοιπόν, εκφράζεται στην τοπική διάλεκτο ο εκπρόσωπος της περιοχής της Ναβάρα. Hasi baino lehen, eskualdetako lantaldea eskertu nahi dut, ekintzailetza arloan Nafarroak egiten duen lana aitortzeagatik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 ekintzailetza plana noski, zientzia teknologia eta berrikuntza plana ere bai, klaster politika, arrisku kapitala, gizarte ekonomiaren osoko plana, ekintzailetzat eta enpresetarako. Let me just interrupt, please. Ζητώ συγγνώμη να σας διακόψω λίγο. Ε, ζητώ συγγνώμη για το γεγονό ότι δεν έχει προβλεφθεί διερμηνία από τα βασικά σήμερα. Επομένως, θα προσπαθήσουμε στο δυνατόν καλύτερα να καταλάβουμε αν δεν, έχετε, αν δεν έχουμε διερμηνία από τα βασικά, λέει ο μιλητή, να συνεχίσω στα καστιλιανικά ισπανικά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή των Περιφερειών, κύριε Αντιπρόεδρε, πρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών ε, αυτοδιοικήσεων, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω ε, δίνοντα τα συγχαρητήριά μου στι άλλε δύο περιφέρειες που βραβεύτηκαν μαζί με εμά και το Κτάνσκ Πομόνσκι και την περιοχή του Κέτεμπερκ. θα ήθελα επίσης να πω ότι το σύστημα της ε, Ναβάρα βασίζεται ε, και μοιάζει με τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει και οι άλλες δύο περιφέρειες. Μέχρι το από το 2016 κάναμε μια αναθεώρηση της στρατηγικής μας για την ευφυή εξειδίκευση και συμμετείχαν σε αυτή εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, τεχνικών, ε, τεχνολογικών Ινστιτούτων, καθώς επίση και εκπρόσωποι της περιφερειακή και της εθνικής κυβέρνησης. Πιστεύω ότι αυτό είναι κρίσιμο, είναι στοιχείο κλειδί. Ε, αυτή η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει ε, και ακριβώς αυτό είναι που έδωσε στο όραμά μας την πνοή και την συνέχεια που χρειάζεται. Στο πλαίσιο της εφιούς εξειδίκευσης και προσπαθώντας να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα, ε, ξεκινήσαμε μια σειρά δράσεων προσπαθούμε να προωθήσουμε την χρήση νέων τεχνολογιών, την, αξιοποίηση των κλάστερ, την αξιοποίηση του, του ενιαίας θηρίδας, έτσι ώστε για να διευκολύνουμε ε, τις επιχειρήσεις. Μικρά βήματα, αλλά αν τα δει κανεί όλα μαζί, δημιούργησαν ένα σύστημα, ένα πλαίσιο επιχειρηματικότητας που ε, φέρνει αποτελέσματα. Αυτό οδήγησε στην συμφωνία της Ναβάρα για την επιχειρηματικότητα. Πιστεύουμε ότι αυτές οι συμφωνίες είναι ε, που δίνουν την ανταγωνιστικότητα στην περιοχή μας. Χρειάζεται κανείς να υπάρξει συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να ενισχύσουμε την καινοτομία σε εκείνους τους τομείς που έχουν ε, εντοπιστεί ως προτεραιότητες στη στρατηγική μας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία ήδη από τη γέννηση της ιδέας του μέχρι την ανάπτυξη της επιχείρησης. Αυτό δημιουργεί μια ευημερία στην περιοχή η οποία βασίζεται και στην επιχειρηματικότητα και στη βιομηχανοποίηση. Ήδη ακούστηκε πώς αξιοποιούμε τις ικανότητες και τα ταλέντα όλων έτσι, και έτσι ώστε η Ναβάρα να διατηρήσει και να βελτιώσει την υψηλή της ανταγωνιστικότητα. Θεωρούμε ότι το βραβείο αυτό είναι μια αναγνώριση των προσπαθειών μας είναι επίσης και μια ενθάρρυνση για να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα έπρεπε να είχαμε και βασκικά ε, ως ε, παθητική γλώσσα. Ε, εν πάση περιπτώσει θα μπορούσατε να έχετε χρησιμοποιήσει τη γλώσσα τη βασκική, αλλά σας ευχαριστούμε για το μήνυμα που μας ε, μεταβιβάσατε. Να κλείσω λέγοντας ότι σας ευχαριστώ όλους σας, όλες ε, τις περιφέρειες που υπέβαλαν ε, υποψηφιότητα αλλά δεν λάβαν το βραβείο. Φέτος αυτές οι τρεις ε, περιφέρειες με τις πόλη σας, με τις βιομηχανίες σας. Θα εργαστείτε σκληρά, θα μας διδάξετε πολλά πράγματα. Είμαι βέβαιο, θα χρησιμοποιήσετε την εμπειρία σας για να αναπτύσσετε περαιτέρω την ε, όλη ιδέα. Και όπως σας είπα θα ανοίξουμε την ετικέτα αυτή της επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικής περιφέρειας ε, για να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Να σας καλέσουμε λοιπόν τώρα σε ένα κοκτέιλ ε, για ένα ποτό μαζί με τους νέους ε, Ευρωπαίους που λάβαν συμμετείχαν στην στο σχετικό διαγωνισμό έξω από το ημικύκλιο. Οι νεαροί λοιπόν Ευρωπαίοι προσκλήθηκαν να μας δείξουν τις φωτογραφικές τους ικανότητες, να βγάλουν μια φωτογραφία που να ενσαρκώνει την Ευρώπη από την περιφέρειά σας. Το ερώτημα ήταν πού και πώς αισθάνεστε την παρουσία της Ευρώπης εκεί που ζείτε. Και επιλέξαμε 20 έργα τα οποία και εκθέτουμε στην αίθουσα που θα λάβει χώρα το κοκτέιλ. Θα σας προσκαλέσω λοιπόν όλους για ένα ποτό. Σας ευχαριστώ πολύ και κυρίσω τη λήξη της σημερινής Ολομέλειας. Να καλέσω και όλους από την πολεμική αντιπροσωπεία και τον Μάρεκ, ο οποίος είναι η οικοδεσπότης της εκδήλωσης στο δικό μας το κτίριο, το κτίριο Jacques Delors. Πέρα τη συνεδρία σα. Ευχαριστώ. Yeah, let's take a photo of...